Δουλεύει, δουλεύει. Uh, Καλησπέρα σε όλους. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο. Παρακαλώ καθίστε όλοι. Θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμα της σημερινής συνεδρίασης, της απογευματινής. Το πρώτο σημείο είναι η γνωμοδότησή μας επί της έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Συγγήτρια, εδώ η κυρία Μπαστός, συντάκτρια της νομοδότησης μάλλον. Να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά, γιατί είναι τα γενέθλιά σας σήμερα, κυρία Μπαστός. Καλώς ήρθατε λοιπόν, ευχές από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Έχουμε λοιπόν την ε, κυρία Μπαστό και ελπίζω και οι σκιώδει να συνεισφέρουν. Η κυρία Βάιλερ ε, σίγουρα είναι εδώ, που να είναι θα έρθει. Ο κύριο Μπουζάη νομίζω θα μιλήσει επίση. Ο κύριο Φόξ είναι εδώ. Ποιο άλλο είναι εδώ ο κύριος Σιντεγκάρντ, Χάιντι θα λάβει το λόγο. Και η ακοπία στην κυρία Ρούλε επίσης. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Σαλβίνη. Τέλος πάντων θα ακούσουμε και τους κοιόδες και τώρα καλώ την κυρία Μπαστός να μας ενημερώσει για τη θέση της σε σχέση με αυτό το σημαντικό σχέ, το θέμα. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και για τις ευγενικές σας ευχές. Επειδή πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν πιο συγκεφαλαιοτική. Ιδίω σε ό,τι αφορά το θέμα της οδηγίας 2001-83, η οποία σκοπό έχει να απαγορεύσει την ε, εισαγωγή των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα της ε, παραγωγής και της κατανάλωσης. Εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα που έχουν παραμείνει εκκρεμοί και παραμένουν εκκρεμοί εξαιτία τη πρόταση τη οδηγία τη Επιτροπή, τα οποία θα ήθελα να παρουσιάσω στου συναδέλφου και να έχω και την γνώμη του. Ένα από τα σημεία αυτά έχει να κάνει με ένα ζήτημα ζωτική σημασία για μα και που έχει φέρει και την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μα το θέμα της δημόσιας υγείας και το συμφέρον του καταναλωτή. Το ενδιαφέρον του να έχει πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία είναι αυθεντικά και δεν θέτουν ε, σε κίνδυνο την υγεία του. Υπ' αυτήν την έννοια υπάρχει προφανής μέρημνα στην πρόταση μεν, αλλά η έκφρασή της στα άρθρα που την αποτελούν ουσιαστικά στέκεται στο φαινόμενο της παραποίησης των ε, φαρμάκων, ένα φαινόμενο με αυξανόμενες διαστάσεις, με μεθόδους όλο και πιο εξελιγμένες και εγκληματικής προέλευσης. Ξέρουμε ότι η αλλαγή της οδηγίας ε, έχει να κάνει με την ε, νομική αλυσίδα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παραποίηση των φαρμάκων είναι ένα μέτρο διάδοσης, χρησιμοποιείται μάλλον ένα μέτρο, μέσο διάδοσης, το ίντερνετ, το οποίο είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν ε, αποτελεί στοιχείο άγνωστο για μας ότι η οδηγία αυτή αφορά το εμπόριο των φαρμάκων, κυρίως το ίντερνετ και δεν μπορούμε να παραμερίσουμε την ε, παραπομπή στη δική μας γνωμοδότηση, την παραπομπή ε, στο ότι το μέσο που κατεξοχήν χρησιμοποιείται από τους παραποιητές των φαρμάκων είναι ακριβώς το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Κάτι άλλο που μας δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την πρόταση έχει να κάνει με την απουσία από την πρόταση ορισμού των ψευδεπιγράφων φαρμάκων. Ο ορισμός αυτός για μας θεωρείται καθοριστική σημασίας, ώστε να γνωρίζουμε επακριβώς ποια ποιο είναι το θέμα το οποίο μας απασχολεί, διότι υπάρχουν κάτι μέλη που γνωρίζουν ότι όταν μιλάμε για ψευδεπίγραφα φάρμακα, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένου όρους, να ξέρουμε τι καλύπτει ο ορισμός δηλαδή. Δεν θέλουμε επίσης να συμβεί κάτι που ήδη συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή να θεωρείται ψευδεπίγραφο ένα φάρμακο από κάποιους και από κάποιους άλλους όχι. Γνωρίζουμε ότι ο ορισμός <clears throat> δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί. Έχουμε όμως και ένα μέτρο στάθμισης. Δηλαδή, ο ορισμός που ακόμη συζητάτε στο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτή η πρόταση στο σχέδιο νομοδότησης πρόκειται να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή θα ήθελα να περάσω σε μια αναδιατύπωση του ορισμού των ψευδεπίγραφων φαρμάκων παραπέμποντας τον ορισμό που έχει χρησιμοποιηθεί και στο επίπεδο του ΠΟΗ. Επίσης, σε σχέση με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των φαρμάκων, εφόσον πρόκειται για ένα φαινόμενο που πλήττει την δημόσια υγεία, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας στα κουτιά των φαρμάκων, ώστε ο τελικός καταναλωτής όλης της αλυσίδας να ε, μπορεί να εξετάσει ενδελεχώς το κατά πόσον τα φάρμακα αυτά είναι αυθεντικά και δεν έχουν υποστεί παραποίηση, παραχάραξη μέσω των διαφόρων δικτύων παραγωγής ως την κατανάλωση. Γι' αυτό σωστά η Επιτροπή κατά την άποψή μας παρουσιάζει προτάσεις για την ασφάλεια και κώδικες συνεννόησης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα στοιχείο μάλλον το οποίο έχουμε αποδεχτεί και σκοπεύουμε τα safety features που θα περιλαμβάνονται στα κουτιά των φαρμάκων, τα στοιχεία ασφάλειας, να καλύπτουν όλα τα φάρμακα ιατρικής, ε, που δίνονται βάσει ιατρικής συνταγής, καθώς και τα καινοτόμα φάρμακα και όσα δεν υπόκεινται σε υποχρέωση ιατρικής συνταγογράφησης. Γνωρίζουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής προχώρησε τόσο πολύ σε ό,τι αφορά τις ε, υποχρεώσεις αυτές, ώστε οι πρακτικές ε, που αποκλίνουν στα διάφορα κράτη-μέλη μεταξύ τους για τα φάρμακα που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση συνταγογράφησης Εφόσον σε μερικά κράτη πολλούνται στα σούπερ μάρκετ τα φάρμακα, ενώ σε άλλα στο, στα φαρμακιά και μόνον. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η πρόταση αυτή έχει σκοπό να προχωρήσει πολύ. Παρά λοιπόν τη δυσκολία και την ανισότητα στη, στο δίκτυο διανομής, δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρο εδώ το θέμα των φαρμάκων που υπόκειται στην υποχρέωση ιατρικής συνταγογράφησης. Επίσης η επανασυσκευασία πρόταση της Επιτροπής εδώ είναι να μην απαγορεύεται η επανασυσκευασία. Όμως εμείς θεωρούμε ότι για να υπάρξει ασφάλεια, πλήρης ασφάλεια, για την δραστηριότητα των parallel traders, των παραλλήλων εμπορευομένων, πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τους ειδικού, τους εμπειρογνώμονες στα θέματα της επανασυσκευασίας. Εδώ δεν έχουμε τελεσίδικη τοποθέτηση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα την τοποθέτηση, των, την άποψη των εμπειρογνωμόνων. Επίσης, θα ήθελα τη συνεισφορά των συναντέλφων για κάποια άλλα στοιχεία, ιδίως για την βασική ημερομηνία, όπως γνωρίζετε για την, για την τράπεζα δεδομένων, ε, θα πρέπει να σεβαστούμε όλους τους κανόνες απόρριτου και εμπιστευτικότητα. <clears throat> και αυτή η βάση θα πρέπει να συσχετιστεί με την παραποίηση των φαρμάκων. Θα την διαχειρίζεται ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ή θα την διαχειρίζεται ένας εθνικός φορέας σε κάθε επίπεδο κράτους μέλους. δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία παραβίαση των πληροφοριών, των κανόνων για την ασφάλεια των πληροφοριών που θα περιέχει αυτή η τράπεζα δεδομένων, βεβαίω. Οι επιθεωρήσεις τώρα είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Οι καλές πρακτικές διανομής πρέπει να ελέγχονται και θα πρέπει να είναι αντικείμενο ελέγχου από επίσημους φορείς. Θα μπορούσε επίσης να υπάρχει συμμετοχή ιδιωτικών φορέων, εταιριών και αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και να ακούσουμε τους ε, ειδικού στον τομέα αυτό. Ιδίως τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους. Για το κόστος, και γι αυτό, με αυτό θα ήθελα να κλείσω, θεωρούμε ότι το κόστος των μέτρων ασφαλείας ως άμεση συνέπεια της υλοποίησης της οδηγίας αυτής θα πρέπει να είναι αναλογικά κατανεμημένα μεταξύ των φορέων της φαρμακοβιομηχανίας και ο τελικός καταναλωτής, ο ασθενής, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί. Δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί στην αγορά και την κατανάλωση φαρμάκων. Σας ευχαριστώ που με προσέξατε την παρέμβασή μου, που μου δώσατε την προσοχή σας και ελπίζω στη, στα σχόλιά σας, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, προκειμένου να ετοιμάσουμε ένα λίγο πολύ επίσημο έγγραφο, ένα σχέδιο γνωμοδότησης ώστε στη συνέχεια με μεγαλύτερη συνέπεια και ακόμη πιο επίσημα να σταθμίσουμε την τοποθέτησή μας για την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστούμε κυρία Μπάστος, μας είπατε τα πιο σημαντικά και όλα αυτά τα οποία είπατε έχουν σημασία για την εσωτερική αγορά στα πλαίσια της αγοράς των φαρμάκων. Τώρα Έχουμε εδώ πέρα τους ασκιούς που ζητήσει το λόγο και πριν του δώσω το λόγο ε, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη που δεν σας παρουσίασα και δεν υποδέχομαι τον κύριο Τέμπεργκερ από την Γενική Διευθυνσία της Κομισιόν για τις επιχειρήσεις. Και έχουμε τους εξή που έχουν ζητήσει τον λόγο. Όλους τους σκιώδεις ηγητές. Ή τους αντικαταστάτες. Mr. Mrs. Ruler, Mr. Fox so far, and Mr. Correa de Campos, uh, so, and Mrs. Steiler. Anybody else? Κανείς άλλος, θέλει το λόγο. Πολύ ωραία. Για τους σοσιαλιστές λοιπόν, κύριε Βάιλερ. Είναι σκιώδης συγκήτρια. sorry, das war jetzt eine falsche Übersetzung. Ναι, ε, η κυρία Στάιλερ είπατε, αλλά τέλο πάντων, εντάξει. Μπα περιπτώσει. Λάθο στο όνομα. Βάιλερ, Στάιλερ, ε, είναι λίγα ίδια τα ονόματα. Κυρία Μπαστό. λυπούμε που θα ακούσετε από μένα κάποιες, ε, μάλλον θα περιμένετε από μένα κάποιες ε, προσθήκες, αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να το κάνω σήμερα σε αυτή τη φάση, γιατί έχετε συμπεριλάβει τόσα πολλά στην δική σας έκθεση που πραγματικά είναι τόσο πλήρης όχι μόνο από την πλευρά της εσωτερικής αγοράς, ξεπεράσατε αυτό το τομέα, οπότε εγώ ήθελα απλώς να σας πω ότι συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Είναι σωστό που λέτε ότι πρέπει να προστατευτούν τα δεδομένα. Είναι σωστό που θίγεται το θέμα των ελέγχων της εποπτείας, Είναι σωστό που θίγεται το θέμα των στοιχείων ασφαλείας mm. Είναι επίση σωστό που Θέλετε να υπάρχει ο ίδιος ορισμός όλα τα ναι. κράτη-μέλη. Και επίσης θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό που λέτε για το κόστος, ότι πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Δεν μπορεί να το μετακυλήσει στους καταναλωτές. Θα δούμε βέβαια πώς θα το διατυπώσουμε στην ε, έκθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει όλα να είναι λογικά και σκόπιμα. Εγώ δεν έχω <coughs> κανένα πρόβλημα με αυτά που προτείνετε στην έκθεσή σα. Απλώ ε, δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Το ένα είναι ε, οι διαφορετικές πρακτικές Θυμάμαι ότι πριν από 10 χρόνια περίπου είχαμε μία περίπτωση με ομοιοπαθητικά προϊόντα και εκεί είχαμε δει ότι είναι τελείως διαφορετική διαχείριση, κυρίως στα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θυμάμαι ότι τότε είχαμε πει δεν το, δεν το βλέπουμε καθόλου αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά θα γίνει επανάσταση αν αρχίσουμε να επιβάλλουμε ό,τι συμβαίνει στη μια χώρα και το, στις υπόλοιπες. Θα δούμε λοιπόν πώς θα το ε, προτείνουμε αυτό στην ε, έκθεσή σας. Και επίσης νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς τώρα να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εναρμόνιση στον τομέα αυτό. Ίσως σε 10-15 χρόνια, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω ότι θα είναι δυνατό αυτό. Και επίσης δεν είμαι σίγουρη για το τι θα γίνει με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ήταν τα πράγματα έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να εξάγει στα, τα υψηλού επίπεδου ποιοτικά προϊόντα της στην Ασία κτλ. Σήμερα δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα πράγματα. Παλαιότερα γινόταν σήμερα όμως όχι. Οπότε θα ήθελα να το ξαναδούμε πώς θα το διατυπώσετε στην έκθεση. Και επίσης, ακριβώς επειδή κάνετε τόσο πλήρη την έκθεσή σας, θα ήθελα εγώ απλώς να επανέλθω στο αίτημα που είχα υποβάλει και μεταξύ των, πρώτης, μεταξύ των ε, σκιωδών εισηγητών για, τις, ε, για την ε, ακρόαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να κάνουμε εμείς κάτι από μόνοι μας γιατί ούτως ή άλλως εμείς ασχολούμαστε περισσότερο με την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές, οπότε νομίζω θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά. Uh, thank uh, Ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Μπουσόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας και συγχαρητήρια για την εισήγηση. Ε, Τώρα χρειάζονται τέτοια μέτρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την νομιμότητα της προσφοράς. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί έτσι η υγεία των ασθενών. Όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί θα πρέπει στην Επιτροπή μα να τα προωθήσουμε. Πρώτα-πρώτα το πεδίο εφαρμογή αυτή τη ανθυρμένη οδηγία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και τα εκτό διαγράφηση ε, φάρμακα. Δεύτερον, να έχουμε κάποιο είδου ε, κριτήρια για τα κριτικά ασφάλεια. Τρίτον, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το παράλληλο εμπόριο και την επανασκευασία και επίση και τη διαχείριση και τον έλεγχο για τη διανομή των ε, φαρμακευτικών προϊόντων με κάποιο είδου νόμιμη αλυσίδα προσφορά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα παραποιημένα Και θα πρέπει όμω να δούμε πώ θα υπάρχει νομιμότητα στην ελευθερία τη προσφορά. Κάτι το οποίο όμω δεν αρκεί, γιατί θα πρέπει να δούμε πώ αυτά τα περιμένα φάρμακα θα τα καταπολεμήσουμε στην Ένωση, γιατί εδώ μιλούμε για οργανωμένο έγκλημα, τέτοιου δραστηριότητα. Η η πρόταση τη Κομισιόν ε, καμιά φορά φαίνεται απονευρωμένη, γιατί το θέμα αυτό παρά είναι σοβαρό όσον αφορά την εσωτερική αγορά και πλευρά καταναλωτών. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να καταπολύσουμε τις παρανομές αγορές, να δυναμώσουμε τα μέτρα προστασίας καταναλωτών από αυτά τα παραπημένα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, πόλη φαρμάκων μέσω του Ιντερνετ. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά, γιατί ε, από εκεί ε, βρίσκουν την κερκόπορτα να μπουν τα παραπημένα φάρμακα. Αυτή πρόταση δεν περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να τη συμπληρώσουμε. Ίσως δεν θα μπορέσουμε όλα τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε τώρα με αυτό το νομοθέτημα. Όμω θα πρέπει αυτή τη συζήτηση να τη χρησιμοποιήσουμε για μια ανοιχτή κουβέντα και να απευθύνουμε έγκριση στην Κομισιόν, τόσο ώστε να μπορέσει να εκπονήσει περαιτέρω πρωτοβουλίε για αυτό το θέμα. Να την ε, πούμε στου ε, καταναλωτέ ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι γίνεται με το Ιντερνετ. Θα πρέπει επίση να δουλέψουμε παραπάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και να προσανατολιστούν σωστά οι καταναλωτέ, οι ασθενεί όσον αφορά τις νόμιμες αλυσίδες προσφοράς, κάτι το οποίο προανέφερα τώρα, αλλά θέλω να σας προσθέσω και κάτι άλλο, ότι αυτή η παραποίηση των φαρμάκων είναι οργανωμένο έγκλημα και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να την καταπολεμήσουμε. Θα πρέπει ε, κάτι να γίνει όσον αφορά το επίπεδο της δικαιοσύνης, τα τελωνία, την αστυνομία, έτσι για αυτά τα φάρμακα. Πέραν της πρώτης αυτήν της Κομισιόν. Έτσι θα κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, ώστε να μπορέσουμε να καταβολήσουμε αυτά τα φάρμακα. Να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη προστασία για τον καταναλωτή και τον ασθενή. Thank σε Εγώ δεν είμαι σκιώδης. Ήμουνα και στη συνάντηση βέβαια εν μέρη παρούσα. Θα συμφωνήσω ε, να ευχηθώ και εγώ στην κυρία Παστό. Ε, χρόνια πολλά. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η ε, έκθεσή της. Υποστηρίζω της, την προσέγγιση της. Θεωρώ ότι όντως είναι σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Γιατί η Κομισιόν αυτό που προτείνει, που προτείνει περιλαμβάνει μόνο 1% του προβλήματος. Το 1% του προβλήματος προκύπτει σε αυτό το νόμιμο δρόμο και το 99% στους υπόλοιπους. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, να πιέσουμε την Κομισιόν. Αν τώρα δεν μπορέσουμε να διευρύνουμε την, αίτηση, την έκθεση, θα πρέπει να κάνουμε μια πρόταση, έτσι ώστε τα θέματα αυτά του ίντερνετ να τα συζητήσουμε ενδελεχώς. Επίσης, ε, να δούμε τι γίνεται με τον ορισμό αυτός, θα πρέπει να είναι η βάση. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε δηλαδή οδηγία. Ε, θεωρώ ότι έχετε προχωρήσει με πολύ σωστό τρόπο. Ε. Και για τα υπόλοιπα σημεία επίσης ε, μόνο να συμφωνήσω μπορώ μαζί σας και βεβαίω να σας προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μας. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και η δική μου ομάδα στηρίζει αυτό το νομοθέτημα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπεζόη. Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί μέρο τη οργανωμένη εγκληματικότητα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα για να αναχαιτήσουμε αυτή τη δράση. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει μια συμπεφωνημένη, ένα συμπεφωνημένο ορισμό. Είναι σημαντικό αυτό για την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση. Να μιλήσω και για το ίντερνετ. Δικό μου φόβο είναι ότι αν τα μέλη αυτή τη επιτροπή προσπαθήσουν να διευρύνουν το πεδίο του νομοθετήματο για να καλύψουμε και το Ιντερνετ, τελικά αυτό που θα πετύχουμε να κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε την έγκριση τη νομοθεσία για πάρα πολύ χρόνο. Εγώ θα προτιμούσα να αφήσουμε τον διακανονισμό των θεμάτων του ίντερνετ σε μια μελλοντική οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό, εάν προσπαθήσουμε τώρα με αυτή την νομοθετική πρόταση να επιλύσουμε και αυτό το θέμα. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει ρήτρα αναθεώρηση σε αυτήν την οδηγία ε, και να το επισημάνουμε αυτό στη γνωμοδότησή μα και για του παράλληλου εμπορευομένου να πω ότι εγώ του στηρίζω και συμφωνώ με τη δράση του γιατί μειώνουν το κόστο για του καταναλωτέ. Για το θέμα του κόστου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τι λύσει που προτείνουμε. Οι λύσει αυτέ να είναι αναλογικέ. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω με την κυρία Μπαστό ότι οι συνταγέ θα πρέπει να καλύπτονται. Απλώς θα πρέπει να πιστούμε ακόμη για το ότι η διεύρυνση της, η, κάλυψη μάλλον των μη συντηγαγραφούμενων φαρμάκων ε, από την οδηγία θα είναι αποτελεσματική. Ιδάλλως ε, νομίζω ότι αν δεν είμαστε προσεκτικοί μπορεί αντί να λύσουμε το πρόβλημα να δημιουργήσουμε περαιτέρω δυσκολίες. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Συνοπτικότατος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε, Αμπάστο, για το έργο το οποίο επετέλεσε πρώτα-πρώτα και που μας τα είπε όλα αυτά σήμερα, σήμερα τη μέρα της γιορτής της. Πάρα πολύ σοβαρά όσα μα ε, ανέπτυξε και να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν σε τέτοια δύσκολα θέματα. Τώρα, παρακάτω. Ανησυχούμε όλοι ιδιαίτερα και με το δίκιο μας για την ε, διάδοση των φαρμάκων μέσω του ίντερνετ. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της πρόληψης της παραποίησης φαρμάκων μέσω του ίντερνετ και να δούμε τι ακριβώς ε, εξουσιοδοτήσεις δίδονται. Και πέραν από τη διευθέτηση του ίντερνετ, και συμφωνώ με την παρέμβαση του συναδέλφου, δεν ε, θα πρέπει τεχνητός να καθυστερήσουμε την πρόταση αυτή και να δημιουργήσουμε δυσκολίες στην έγκρισή τη, προσπαθώντας να διευθετήσουμε και το ίντερνετ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν η Επιτροπή έχει υποβάλει την πρόταση αυτή σε ένα φαρμακευτικό πακέτο, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αλλαγή στον, ε, στην οδηγία και τους κανόνες σε σχέση με την πληροφόρηση, την ενημέρωση των καταναλωτών. Ο καλύτερος τρόπος να διαθετήσουμε το ίντερνετ και να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείται ορθώς είναι τα φάρμακα που διαθέτονται μέσω του ίντερνετ να παρέχουν ε, απαραίτητες εγγυήσεις. Δεν είμαι υπεραισιόδοξος λέγοντας ότι καλή ενημέρωση θα αποβάλει από το ίντερνετ ουσιαστικά με τρόπο φυσικό τα φάρμακα που δεν είναι κατάλληλα. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε για την καλή ενημέρωση έστω και μέσω του ίντερνετ. Αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να το πετύχει η οδηγία για την... η παράλληλη οδηγία για την... Ε, και ο κανονισμός για την ενημέρωση των ασθενών. Θα συμφωνήσω επίσης με τον συνάδελφο Fox διότι και εγώ ακόμη απομένει να πιστώ για τα θέματα ασφάλειας και για το πώς, κατά πόσο μπορούμε να καλύψουμε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Θα πρέπει να ενισχυθούμε λοιπόν, να ενισχύσουμε εδώ τους κανόνες ακόμη και για τα συνταγογραφούμενα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα επικουρικότητας, διότι υπάρχουν χώρες που έχουν μεθόδους πώληση και διανομής των φαρμάκων, τα οποία μοιράζονται και συσκευάζονται σε φαρμακεία, ενώ Υπάρχει και η βιομηχανία που δεν αποδέχεται τον κατακαιρματισμό της ε, πώληση στα φαρμακεία με μεθόδους ασαφείς και άγνωστες κάποιες φορές Κάτι που είναι δικαιολογημένο για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, αλλά όχι για τα μη συνταγογραφούμενα. Εδώ νομίζω ότι αν αλλάξουμε αυτούς τους κανόνες θα επιφέρουμε πρόσθετο κόστος. Και τα, τα φάρμακα αυτά πολλές φορές είναι γενώσιμα, οπότε θα επηρεαστεί σαφώ το κόστος τους. Θα πρέπει λοιπόν ο στόχος της Επιτροπής μας είναι να, να είναι να διευκολύνουμε τους καταναλωτές ε, επίσης, ένα τελευταίο σχόλιο. Όλοι θα θέλαμε ο κόστος των, το κόστος των μέτρων ασφαλεία να μην επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Όλοι αυτό θέλουμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε τουλάχιστον εν μέρη ένα, ένα μέρος από το κόστος αυτό να επιβαρύνει όντως τους καταναλωτέ. Η μόνη εναλλακτική που μένει είναι τα κόστη αυτά να βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον παραγωγό. Εφόσον ε, υπάρχουν ε, διάφοροι φορείς όμως στην αλυσίδα παραγωγής, ε, σε πολλα κατημέλη που αμείβονται βάσει του αρχικού κόστους του προϊόντος, του φαρμάκου. Η ευχή αυτή λοιπόν, η επιθυμία αυτή είναι αξιοσέβαστη θα έλεγα, ιδιαίτερα αξιέπαινη, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτέ ήταν οι δικέ μου γενικέ παρατηρήσει. Είμαι βέβαιο ότι η συνάδελφο Ρεζίνα Μπάστου θα τα λάβει υπόψη. Ευχαριστώ. Uh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και χρόνια τους πολλά. Πολλά από όσα υπόθηκαν τα υποστηρίζω και εγώ. Το θέμα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, είναι ένα θέμα σημαντικό. Είναι παράνομα και μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και θάνατο στους καταναλωτές. Και μπορεί οι καταναλωτές να παραπλανηθούν και να αγοράσουν κάτι που να είναι όντως ψευδεπίγραφο. Πραγματικά λοιπόν η ευθύνη μας είναι μεγάλη για να δούμε το θέμα αυτό. Και η συγγήτρια το έχει τονίσει στην έκθεσή της και είναι στη σωστή χρονική στιγμή επίσης. Η κυρία Βάιλερ μίλησε για την οδηγία για, τις, για τα ομοιοποθετικά φάρμακα. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ ως προς αυτό, αλλά αυτοί που παράγουν αυτά τα φάρμακα παράγουν ένα ποιοτικό προϊόν. Βρίσκεται όμως στην αγορά κάποια πράγματα τα οποία ε, κατά 75% αποτελούνται από στάχτη. Είναι δηλαδή σοκαριστικό το να σκεφτεί κανείς τι αγοράζει τελικά ο καταναλωτής. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα ομοιοπαθητικά προϊόντα που μπορεί να αγοράσει. Όπως είπε και ο κύριος ε, Κάμπος, για τις διαφορετικές παραδόσεις που έχουμε στα κράτη-μέλη, στην οδηγία για τα πρόσθετες ουσίες στα τρόφιμα. Είδαμε ότι όντως υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές στα κράτη-μέλη και πρέπει όντως να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της ε, επιλογής του καταναλωτή και της ασφάλειας. Οπότε και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Για το ίντερνετ τώρα και τα όσα το αφορούν πολλοί καταναλωτέ όντω αγοράζουν από το ίντερνετ και θα με ενδιαφέρει να ακούσω από την Κομισιόν ποια, πόσα μάλλον ψευδεπίγραφα φάρμακα ε, αγοράζονται από το ίντερνετ και αν υπάρχουν σχετικέ πληροφορίε. Στη δική μου την εκλογική περιφέρεια, να σα πω, το, ποσό, το ποσοστό των ανθρώπων που ε, εθίστηκαν σε προϊόντα μαυρίσματο που αγόραζαν από το ίντερνετ, που ήταν παράνομα αλλά μπορούσαν να τα βρουν στο ίντερνετ, ήταν, έκαναν ενέσεις για να μαυρίσουν, ήταν πραγματικά σοκαριστικό και ε, εθίστηκε ο κόσμος αυτός. Και δεν νομίζω καν ότι αυτά τα φάρμακα έχουν ε, τύχη και της σωστής, ε, του σωστού χαρακτηρισμού. Και πολλοί γιατροί το έθιξαν το θέμα αυτό. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Φόξ για τα φάρμακα με, χωρίς συνταγογράφηση, θα πρέπει να δούμε αν είχε γίνει η αξιολόγηση επιπτώσεων για τα συγκεκριμένα φάρμακα γιατί πραγματικά κατανοώ αυτά που λέει και ο κύριος Κάμπος και ο κύριος Φόξ. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. μην ε, ε, τρομάζετε πολύ από τα από τα προϊόντα μαυρίσματο, ε, αλλά πραγματικά εγώ σοκαρίστηκα όταν το έμαθα. Δεν το χρησιμοποιώ βεβαίω, αλλά πραγματικά τρομοκρατήθηκα μόλι έμαθα για αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ που προσθέσατε μια νέα διάσταση στη συζήτησή μα. Η κυρία Σαρτόρη επίσης εισηγήτρια συγγνώμη, για τα βιοκτώνα. Είναι το τρίτο σημείο που θα δούμε αύριο. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει και την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων της για τα βιοκτώνα, οπότε θα το δούμε αύριο αυτό. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και αυτό φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλό και για τη δουλειά που έχει κάνει η κυρία Μπάστος. Είναι πολύ σημαντική η διατήρηση των σχέσεων με, τις, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ παρούσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζήτησα να παρέμβω, διότι είμαι εισηγήτρια στην Επιτροπή Βιομηχανία για την οδηγία αυτή, την πρόταση οδηγία. Ήθελα να επιβεβαιώσω και στη δική σας επιτροπή ότι η κατεύθυνση που ακολουθεί η κυρία Μπάστους είναι αυτή που ακολουθώ λίγο πολύ και εγώ ως εισηγήτρια της Επιτροπής Βιομηχανίας. Θεωρώ ωστόσο ότι πρέπει να κάνω δύο σημαντικές διευκρινήσεις σε αυτή τη φάση. Η πρώτη είναι ότι μιλάμε για φάρμακα προϊόν που διαφέρει από όλα τα άλλα. Από οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Εδώ μιλάμε για τη θεραπεία ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίε. Όταν μιλάμε λοιπόν για φάρμακα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ε, ανησυχούμε λιγότερο για το κόστος της δράσης που προτείνουμε και περισσότερο για την εγγύηση, την πλήρη προστασία που μπορούμε να εξασφαλίσουμε, την πλήρη ασφάλεια που πρέπει να περιλαμβάνει το προϊόν αυτό για τον οποιοδήποτε χρήστη. Όποιο χρησιμοποιεί λοιπόν ένα φάρμακο θα πρέπει να αισθάνεται απολύτω προστατευμένο, απολύτω ασφαλή. Έπειτα όλα τα υπόλοιπα έπονται. Εδώ είναι δύσκολο να πετύχουμε το στόχο αυτό, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν δύο διαφορετικέ οδοί που μπορεί κανεί να ακολουθήσει. Πρώτα απ' όλα η χνηλασιμότητα, η πλήρη χνηλασιμότητα, είτε στην αλυσίδα παραγωγή όλων, με όλες τις, τις συνιστώσεις, είτε στην αλυσίδα πώληση με όλες τις, τις συνιστώσεις επίσης και, όλες τις, και όλα τα πλοκάμια. Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να ακολουθήσουμε και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα, διότι ε, τα χρονικά διαστήματα που μας προτείνει η Επιτροπή για να προβλέψουμε ασφάλειες ορισμένα από αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σύντομα θα πρέπει λοιπόν να δικαιολογήσουμε τις προτάσεις μας. Ε, υπάρχει ένα αδύναμο σημείο συγκεκριμένα, αυτό που αφορά τις ενεργές ουσίες. Γνωρίζουμε ότι σε ένα φάρμακο εν τέλει αυτό που πραγματικά μετράει είναι οι ενεργές ουσίες, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία. Τα συνθετικά λοιπόν τα ενεργά είναι ένα στοιχείο αδυναμίας της πρότασης, διότι η πρόταση της Επιτροπής μιλά ακόμη για δύο δυνατότητες, δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτοί των χωρών που παράγουν και αποτελούν μέρος ενός καταλόγου κρατών που μπορούν να μας διασφαλίσουν, να μας ε, καθησυχάσουν και αυτών που περιλαμβάνονται σε ένα κατάλογο παραγωγών χωρών, κρατών που δεν μπορούν να μας παρέσχουν τις απαραίτητες ε, εγγύησεις. Θεωρούμε ότι ο χρόνος της τριετίας που προβλέπεται πριν από την παρέμβαση είναι υπερβολικά μεγάλος. Όμως, <clears throat> θέλω να πω και στη δική σας επιτροπή για του εσωτερικού εμπορίου, κάτι που θα επαναλάβω και στην Επιτροπή Βιομηχανίας, ότι όπου υπάρχουν δυσκολίες για την αποδοχή των επιβλέψεων και των επιθεωρήσεων των μηχανικών ε, των ε, σημείων παραγωγής μάλλον, των βιομηχανιών, αυτό είναι περίεργο, διότι υπάρχουν χώρες όπως οι ΗΠΑ και αλλού που αυτό το πρόβλημα έχει επιληθεί μιας διαπαντός δεν έχει παύσει η παραγωγή, ούτε έχει καθυστερήσει, γιατί υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης και επιθεώρησης των ε, εργοστασίων παραγωγής. Εμείς λέμε ότι είναι δύσκολο, περίπλοκο, γιατί λόγω χάρη, για, για, για τις ενεργές ουσίες υπάρχουν τουλάχιστον 20 εξωτερικά σημεία παραγωγής που παρέχουν ε, τα στοιχεία αυτά στην Ευρώπη. Όχι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Η Επιτροπή λέγοντας κάτι τέτοιο γνωρίζει ότι ο κόσμος και τη κοφιντούστρια και άλλων χωρών μας εξηγούν ότι οι ενεργές ουσίες ε, στο εξωτερικό δεν ξεπερνούν τα σημεία που παράγονται τα σημεία που παράγονται τα πέντε στον αριθμό. Ακόμη και αν είναι 520.000 τα σημεία αυτά, εμείς θα πρέπει να τα, ε, να τα επιθεωρούμε. Να μπορούμε να τα ελέγξουμε ανα πάσα στιγμή. Γιατί οι ενεργές ουσίες βρίσκονται στην ρίζα της θεραπείας οποιασδήποτε ασθένειας ούτως ή άλλως. Θέλετε να παρέμβετε. Εγώ πήρα μοτίλιουμ σήμερα το πρωί που δεν χρειάζεται συναστεγογράφηση ε, και αισθάνομαι καλύτερα. Αλλά αν ε, ήξερα ότι είναι ψευδεπίγραφο το φάρμακο, δεν θα μπορούσα εδώ να μιλώ <coughs> εκ μέρους της κυρίας Πρεβάνοβα, που είναι στην ομάδα γυναικών. Τα ψευδεπίγραφα πραγματικά μπορεί να δημιουργήσουν ε, τραγικά προβλήματα στους καταναλωτές. Yes. Okay. Um, uh, uh, Ως πρόεδρος να κάνω κι εγώ δύο-τρεις παρατηρήσεις. για το ίντερνετ και τις πωλήσει μέσω ίντερνετ. Θα πρέπει να θυμόμαστε, και το λέω αυτό στον ε, κύριο Μπουσόη, ο οποίος κουβεντιάζει κιόλα, ότι είναι ένας τρόπος για να σας πω ότι η πρόταση που δουλέψαμε, επί της οποίας δουλέψαμε εμείς, για, τα, για την οδηγία για τα δικαιώματα των, ε, των καταναλωτών συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα και θα αρχίσει να θα τεθεί σε ισχύ άμεσα. Και αυτό πραγματικά χαίρομαι πολύ που συνέβη και ευγνωμονώ του συναδέλφου. Αλλά σε αυτή την πρόταση περιλαμβάνεται κάτι που έχει συντάξει δική μα επιτροπή, που είναι η δυνατότητα οι ρυθμιστέ των, ηλεκτρονικών, των συστημάτων ηλεκτρονική ε, επικοινωνία να ζητούν, να έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους παρόχους να, να δίνουν μηνύματα ε, σε όλους τους, να στέλνουν μηνύματα σε όλου τους ε, καταναλωτές. Εγώ όταν, όταν συζητούμε την διάταξη αυτή χρησιμοποιώ ακριβώς αυτό το ζήτημα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και τη δυνατότητα να στέλνουμε προειδοποιήσεις στους καταναλωτές για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν να παρουσιαστεί στην υγεία τους. Ε, όταν αγοράζουν τέτοιου είδου φάρμακα, ψευδεπίγραφα. Και αυτό το χρησιμοποιώ ως καλό παράδειγμα για το γιατί είναι σημαντικό να έχουμε αυτή τη διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται τώρα στον κανονισμό, για τη δημόσια ασφάλεια. Ίσως η κυρία Μπαστός λοιπόν θα μπορούσε να το συνδέσει και αυτό, γιατί αυτή είναι νέα διάταξη που υπάρχει, οπότε ίσω θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε. Και επίση αυτό σχετίζεται και με το όλο θέμα τη ασφάλεια, τη συσκευασία, γιατί αν ο καταναλωτής έχει <coughs> τις ε, πληροφορίες και ξέρει τι πρέπει να ψάξει έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι τα στοιχεία ασφάλειας υπάρχουν και είναι ασφαλή ε, ε, η συσκευασία και δεν έχει ανοιχτεί το φάρμακο από το ίντερνετ, αυτό όντω προσφέρει στην ασφάλεια. Γιατί Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα που αφορούν, που απασχολούν τους καταναλωτές πολύ αγοράζουν ε, φάρμακα από τα οποία εξαρτώνται, ας πούμε, φάρμακα ενάντια ε, στην κατάθλιψη. Ε, και πολλές φορές έχουν προβλήματα διότι δεν παίρνουν τελικά, δεν φτάνουν στα χέρια τους τα φάρμακα που θεωρούσαν ότι έχουν αγοράσει. Μου φαίνεται λοιπόν ότι για να προχωρήσουμε και για να είμαστε και αρκετά ρεαλιστές ώστε να είναι και αποτελεσματικό, το πρώτο βήμα θα πρέπει όντως να αφορά τα ε, φάρμακα με συνταγογράφηση. Καταρχήν γιατί είναι πολύ πιο προφανής η κίνδυνη και δεύτερον γιατί το περιθώριο κέρδους που υπάρχει για άτομα που πουλούν τέτοια ψευδεπίγραφα ή παράγουν ψευδεπίγραφα φάρμακα και δεν δίνουν καμία πληροφόρηση από αυτού, είναι πραγματικά πολύ υψηλό το ποσοστό όλων αυτών, γιατί αυτά θεωρούνται και τα πιο αποτελεσματικά υποτίθεται. Και περιλαμβάνουν υποτίθεται τα πιο ακριβά συστατικά. Και εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο κέρδους. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όντω έτσι να προχωρήσουμε πιο στοχοθετημένα. Και επίση, η διαθεσιμότητα είναι πολύ σημαντική. Η διαθεσιμότητα των, ε, των πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες ε, στο φύλλο οδηγιών των, φαρμα, των φαρμάκων. Η παράλληλη διανομής είναι οι, κάποιοι από τους παράλληλου διανομής όντως λειτουργούν ε, κάτω από συγκεκριμένα πρότυπα ε, και λειτουργούν πολύ σωστά, αλλά πραγματικά δαπανούν πάρα πολλά χρήματα στην ανασυσκευασία και στην ε, ετικετοθεσία εκ νέου. Και το τελευταίο σχόλιο που ήθελα να κάνω για την Επιτροπή μας είναι ότι όντω έχουμε κάνει πολλή δουλειά στην Επιτροπή αυτή για την αξιολόγηση και τους, την εποπτεία. Πολλά τα κάναμε για την αμοιβαία αναγνώριση των ε, διαφόρων αγαθών. Και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και στον τομέα της, ε, των φαρμάκων. Νομίζω λοιπόν ότι η κυρία Μπαστός έχει πραγματικά την εμπειρογνωμοσύνη για να τα, συνδυάσει όλα αυτά. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ε, επιπροσθέμενη προσθέμενη αξία που μπορεί να φέρει η δική μας νομοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η κυρία Σαρτόρη επίσης είναι εδώ, οπότε πρέπει όντως ε, να προσθέσουμε στην γνωμοδότηση. Αυτά από μένα. Τώρα, να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Τίερμπεργκερ για να μας πει τη δική του άποψη και μετά θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Μπαστός για να κλείσουμε τη συζήτηση επ' αυτού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. αφού μου δίνετε την ευκαιρία να σας σχολιάσω κάποια από τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Πρώτα πρώτα να τονίσω ότι ευχαριστούμε για τη συνεργασία, για την κατανόηση του πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα αυτών των παραπημένων των ψευδεπήρεγων φαρμάκων. Επίγει το να θεσπιστεί αυτό το νομοθέτημα. και να μπορέσει να διεκπληρωθεί αυτό το ζήτημα στα πλαίσια των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Και επιτέλου να έχουμε κάποιο πιο αυστηρή νομοθεσία, τόσο να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Σύντομα, τώρα όσον αφορά κάποια από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ, διότι τα πιο σημαντικά ζητήματα αφορούν την νομοθετική πρόταση. Και κατά πόσον εμείς είχαμε το, το, το, το, το δέον εύρος στην πρότασή μας καλύψαμε όλα τα θέματα αυτά που τώρα όσον αφορά τις πωλήσει μέσω του ίντερνετ όπως σωστά ε, αναφέρθηκε έγινε αυτή η πρόταση επί της οποίας θα πρέπει να σας πω ότι λόγω των, της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους αλλού επιτρέπεται τέτοιο εμπόριο και αλλού όχι. Οπότε δεν μπορούσαμε να επισέλθουμε για αυτό το λόγο σε αυτό το θέμα. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται περί παρανόμων ιονίων φαρμακείων που πολλούν μέσω του ίντερνετ. Έχουμε επομένω όλου αυτού του παράνομα εμπορευόμενου στο Ιντερνετ. Επομένω αυτό είναι θέμα απλώ εφαρμογή του νόμου. Πρόσφατα, κάποιο κρατοσμένος μας είπε ότι άρχισε ένα πιλωτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο προσπαθεί να έρθει σε επαφή με αυτούς τους πολιτές και να τους πει να το σταματήσουν. Άρα θα πρέπει τώρα να κάτσουμε και να κάνουμε διαχωρισμό. Από τη μία μεριά είναι τα θέματα της εφαρμογής του νόμου και από την άλλη μεριά είναι τα θέματα τα νομοθετικά. Όμως ε, δεν είμαστε εμείς κατά. αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ε, περιθώριο ε, προσθήκης τέτοιου είδους στην πρότασή μας, να το, να το δούμε. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να σεβαστούμε τις ε, εθνικές αρμοδιότητες. Επίσης, επίσης όσον αφορά το παιδί εφαρμογής οδηγίας, έχουμε τα θέματα των ορισμών. Που ε, και, και πάνω σε αυτό μας επικρίνεται και στο Συμβούλιο μας επέκριναν. Θεωρούμε σημαντικό ότι ο ορισμός και στα ψευδεπίγραφα φάρμακα θέλουμε να αποφύγουμε να μπούμε στα χωράφια της πνευματικής διοκτησίας. Πάνω σε αυτό δουλεύει άλλωστε και η Task Force του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και ας μην έχει επιδοθεί ακόμα συμφωνία και συνεχίζουν. Τώρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλεια. θα πρέπει στα σοβαρά να λεφθεί υπόψη το κατά πόσον αυτά τα φάρμακα Πολύ, πολύ σοβαρά λοιπόν λύσαμε το θέμα όσον αφορά αυτό το φάρμακο χωρί συνταγογράφηση για το αν θα καλυφθούν ή όχι. Και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει ο ίδιο βαθμό κινδύνου όπω για τα φάρμακα κατόπιν συνταγογράφηση. Επίσης, οι παρενέργειε αυτών των φαρμάκων των χωρί συνταγογράφηση και αυτές ε, ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο. Φυσικά και δεν υπάρχει μηδενικό κίνδυνο αλλά πολλέ φορέ εδώ έχουμε διαφορετικούς διάβλους ε, διανομής, καμιά φορά διανέμονται αυτά και από το σούπερ μάρκετ. Άρα, είπαμε να περιοριστούμε στα φάρμακα τα οποία χορηγούνται κατόπιν συνταγή. Ε, Επίση, έχουμε τώρα θέμα το τι θα γίνει με αυτά τα χαρακτηριστικά τη ασφάλεια και τι τεχνολογικέ λύσει θα επιλεγούν. Οπότε, και εδώ υπήρξε και το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό είπαμε να προσέξουμε η νομοθετική μας πρόταση να, να, να, να, να κάτσουμε και να δούμε κατά πόσο θα έχουμε μια τέτοια τεράστια τράπεζα δεδομένων και κατά πόσο θα μπορούσαμε να καταγράψουμε και τα πάντα. Αλλά και αυτό ε, αποτελεί κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα. Επομένως και αυτό το αφήσαμε έξω την πρόταση. Αποφύγαμε και αυτό το όλη στήρο μονοπάτι. Όσον αφορά τώρα την συνεργασία των διαφορετικών αρχών και φορέων, εδώ τονίζουμε ότι είναι γεγονός η συνεργασία, υπάρχει. Εδώ και ένα χρόνο. Προβλέπεται, ε, συνομιλούν οι επικεφαλής των ε, φαρμακευτικών οργανισμών κάθε κράτους, συνεργάζονται και με την ε, αστυνομία. Επομένως, το θέμα αυτό έχει πάρει το δρόμο του ούτω ώστε να μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίε και να μπορούμε να συγκεράσουμε τη δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης τώρα τελεί διαπραγματεύσεις όσον αφορά κάποια θέματα ποινικού δικαίου για την παραποίηση φαρμακών. Και αυτό σημαντικό. τελευταίο και σημαντικό. Για αυτά τα, τα στοιχεία που, που περιέχονται στα φάρμακα υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια μηχανίες. Πρέπει να γίνει συνεργασία και εδώ όλων των εμπλεκομένων αρχών, να συνεργαστούμε με όλε τι χώρε οι οποίε εξάγουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα ενεργά συστατικά. Συγκεκριμένα είναι η Κίνα και η Ινδία. Ήδη έχουμε αρχίσει συνομιλίε με αυτέ τι χώρε. Άμεσε συνομιλίε, τόσο ώστε να μπορέσουμε να συντάμουμε την ε, μεταβατική περίοδο και να κάνουμε κάτι για το θέμα που μα ενδιαφέρει η κυρία Σαρτόρια να έχουμε κάποιες εγγυήσεις από αυτές τις τρίτες χώρες. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να δουν σοβαρά το θέμα. Και να κάνουν κάτι για αυτές τις βιομηχανίες οι οποίες ε, εξάγουν προς την Ευρώπη. Να ασχοληθούν οι διοκτικές αρχές των χωρών αυτών. Menschen Τελευταίο αλλά σημαντικό, σας αναφέρω το ότι έχουμε και κάποια ευθύνη ως ε, εξαγωγής φαρμάκων. Γιατί πρέπει να προσέξουμε και τα θέματα τη ε, ποιότητα. Ήδη προβλέπονται κάποιε διατάξει. Δεν πρέπει ποτέ να εξαγάγουμε κάτι το οποίο να είναι κατώτερο των, ε, των προτύπων που έχουμε επιβάλει για μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για τον χρόνο σα. Well, thank Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που καλύψατε τόσα διαφορετικά σημεία. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάστους για να ανακεφαλαιώσει και να μας δώσει και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για το πώς θα προχωρήσει η εξέταση του θέματος. Κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές, τους συναδέλφους που έδωσαν τις ιδέες τους και τη συνεισφορά τους για το ζήτημα αυτό που είναι τόσο ευαίσθητο. Επίσης να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις διευκρινήσεις που μόλις μας έδωσε. Σε ό,τι αφορά σημεία κλειδιά, καθοριστικά σημεία που τέθηκαν, για τη δική μου την εργασία είναι σημαντικό να γνωρίζω ότι κάποια σημεία θα έχουν αποσαφινιστεί πλήρως και θεωρούνται σημεία συμφωνίας για όλους, όπως συγκεκριμένα η ανάγκη για τον ορισμό, το ζήτημα των ενεργών ουσιών και πέραν των όσων είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάγκη αναγνώρισης, αμοιβές αναγνώρισης μεταξύ των χωρών και όσο το δυνατόν πιο σύντομα για τις ενεργές αυτές ουσίες, τα ενεργά συστατικά και εδώ να ευχαριστήσω και για τη συμβολή σας σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή αυτής της αναθεώρησης οδηγίας. Ω προς αυτό, σωστά υπόθηκε και κατέστη εδώ σαφέ ότι όλοι ε, ορμώνται από την ίδια μέρημνα, δηλαδή να γνωρίζουν να διαθετήσουμε και την πώληση ψηφιακών φαρμάκων μέσω ίντερνετ. Ε, μα είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρο τη Επιτροπή μα ότι εδώ υπάρχει συσχετισμός με τις οδηγίες που εγκρίθηκαν και γι' αυτό θέλω να συγχωρώ τον πρόεδρο κύριο Χάρμπορ για το πακέτο Telecom και αυτό ίσως είναι ένας έμεσος τρόπος να διευκολύνουμε το έργο μας εδώ. Δηλαδή, η χρήση του ίντερνετ από τους καταναλωτές να διέπεται και από τους κανόνες των άλλων οδηγιών και να πλαισιώσουμε σωστά και την πώληση φαρμάκων μέσω αυτού του τεχνολογικού μέσου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συνεισφορά είναι σημαντική και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει αντιρρήσεις στο να καλύψουμε με το πεδίο εφαρμογής και τις υπόλοιπες κατηγορίες όπως έχουν οριστεί στην πρόταση οδηγίας. Για τα φάρμακα χωρί συνταγογράφηση, μάλλον έχουμε διαφορετικέ απόψει. Θα πρέπει να τι σταθμίσουμε καλύτερα, διότι όλε οι παρατηρήσει που ακούστηκαν εδώ αξίζουν την ιδιαίτερη προσοχή του. Πρέπει να μελετήσουμε λοιπόν όλες τις απόψεις και να τις αναλύσουμε προκειμένου να αποφανθούμε. Γνωρίζουμε ότι το να εισάγουμε και αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων και τους ίδιους μηχανισμούς ασφαλείας για αυτά όπως είπε και η κυρία Σαρτόρη, είναι σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη προστασία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το ανάλογο κόστος. Το κόστος αυτό δεν πρέπει να είναι υπέρμοτρο και να μετριαστεί το πλεονέκτημα που μπορεί να μας φέρουν τα φάρμακα αυτά. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα φάρμακα, τα όταν τα λαμβάνει ο τελικό καταναλωτή, μπορεί να έχουν σοβαρέ παρενέργειε στην υγεία του. Είναι λοιπόν αυτό η βασικότερη μα μέρημνα. Σε κάθε περίπτωση, σε καθόλου δεν είναι ε, σημαντικό να μετά από μια μελέτη αντικτύπου που δεν έχει γίνει ακόμα και θα πρέπει να είναι λεπτομερής να αποφανθούμε πλήρως για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ιδίω ό,τι αφορά τα φάρμακα που πολλούνται ελεύθερα και αφήνοντα κατά μέρο τις μεθόδου εμπορία των φαρμάκων αυτών στα διάφορα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, να πω ότι η δική μα βασική ε, ανησυχία να υπάρχει ισότιμη κατανομή του κόστους μέσω της οδηγίας είναι πάντοτε η πιο σημαντική, όπως είπε και η συγκήτρια Σαρτόρη. Πιο σημαντικό και από το κόστος είναι η ασφάλεια των ασθενών. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι η δική μας η παραγωγή φαρμάκων έχουν επί της ουσίας συμφέρον η ασφάλεια αυτή να παρασχεθεί. Εφόσον η παραποίηση φαρμάκων είναι και δραστηριότητα που ε, θίγει την φαρμακοβιομηχανία και με τρόπο ιδιαίτερα σοβαρό. Τα κόστη που αυτή τη στιγμή επομίζονται οι επιχειρήσεις λόγω της παραπίσης των φαρμάκων ίσως να αντισταθμιστούν εάν υπάρξει ένα εργαλείο το οποίο να το καλύπτει από την άποψη του κόστου η ίδια φαρμακοβιομηχανία αλλά τα φάρμακα να έχουν πλέον μηχανισμούς που να εγγυώνται την ασφάλεια και την αυθεντικότητά τους. Πρέπει να ευχαριστήσω για τις συνεισφορές σας, οι οποίες ήταν όλες ιδιαίτερα επικοδομητικές και να πω ότι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε, αυτό που έχω στα χέρια μου, θα πρέπει έτσι περαιτέρω να διευκρινιστεί. Η κυρία Μαρίζα Ματίας είναι η επί της ουσίας αρμόδια εισηγήτρια. Έπειτα το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην Επιτροπή ΕΜΒΙ τον Απρίλιο και τότε θα εγκριθεί η έκθεση αυτή και θα ψηφιστεί τον Μάιο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Okay, well, thank you very much indeed, uh, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Μπάστος. δώσατε και τη μισή σας μέρα από τα γενέθλιά σας για να είστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ξεκόραση και καλά να περάσετε από εδώ και μπρος. Λοιπόν, περνούμε στο επόμενο σημείο. Πολύ σημαντικό και πολύ ενημερωτικό. Θα ακούσατε από τη συζήτησή μας και το πρωί και σήμερα τώρα το απόγευμα για τα θέματα επιβολής του νόμου. Μάλιστα κυρίως στον τομέα της ε, προστασίας των καταναλωτών. Το 2004 η Επιτροπή αυτή ήταν υπεύθυνη για την έγκριση του πρώτου κανονισμού για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνε για την επιβολή του νόμου που αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η συγγήτρια ήταν η κυρία Γκέπχαρτ τότε η οποία βεβαίως ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το πώς εξελίχθηκε αυτός ο κανονισμός και πώς εφαρμόστηκε. Η Κομισιόν έχει υποβάλει δύο εκθέσεις, δημοσιεύθηκαν στις 2 Ιουλίου, σε σχέση με τη λειτουργία αυτής της οδηγίας κανονισμού, του κανονισμού για τον οποίο ήταν υπεύθυνη η κυρία Γκέπχαρτ και για κάποιες άλλες πτυχές από των οποίων εργάζεται η Κομισιόν για την εφαρμογή του κεκτημένου των καταναλωτών. Πρέπει να έχετε στους φακέλους σας μια περίληψη για μία από αυτές τις δράσεις. Ε, ζήτησα από την κυρία Κούναβα την προηγούμενη εβδομάδα όταν με προσκάλεσαν για, την, ε, για τον εορτασμό των 10 χρόνων της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ. Ε, έχει εισαγάγει ένα νέο όρο, τον όρο SWEEP, όσοι παρακολουθείτε την δουλειά της Κομισιόν επ' αυτού, θα έχετε δει την ε, που γίνεται και online και στο ίντερνετ, ε, αυτός ο όρος θα αφήσει μάλλον εποχή στην Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Αυτό λοιπόν που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε την Κομισιόν, ο κύριος Τάμας Μόλναρ που είναι, υπεύθυν, είναι ε, επικεφαλής της ε, μονάδας για την των καταναλωτών είναι εδώ για να μας κάνει παρουσίαση και βεβαίω να απαντήσει στι ερωτήσει εφόσον υπάρξουν ε, για τι δύο αυτέ εκθέσει. Χαίρομαι λοιπόν πολύ. Καλώ ορίσατε στην Επιτροπή μα. Πρέπει να υπάρχουν οι διαφάνειέ σα. Υπάρχουν και ε, αντίτυπα, αλλά είναι. Πρέπει να βλέπετε τις οθόνες και τις διαφάνειες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τα απορίσματα και μετά όποιος θέλει να πάρει το λόγο, ευχαρίστως να τον ακούσουμε θα τολμήσω να βάλω την κυρία Γκέπχαρτ πρώτη-πρώτη στον κατάλογό μου και μετά θα ακολουθήσουν και όσοι άλλοι το επιθυμούν. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much for the invitation. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα δύο αυτά έγγραφα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Όντως, όπως είπατε, η εφαρμογή βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής για τους καταναλωτές. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα διαφάνειες. Εν πάση περιπτώσει, όπω είπατε λοιπόν, η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική γιατί θεωρούμε στη ΣΑΝΚΟ ότι δεν, είναι, δεν αρκεί να δώσουμε τα δικαιώματα στου ε, πολίτε μα. Πρέπει να εξασκούνται τα δικαιώματα αυτά και να εφαρμόζονται. Όταν μιλούμε για τι αξίε τη Ευρώπη, μιλούμε για το ότι ίσως να έχουμε πολλούς κανόνες και να μην τους ακολουθούμε. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες ε, εφαρμόζονται. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και γι' αυτό πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή, στην καλύτερη εφαρμογή και γι' αυτό μας προέκυψε αυτό το πακέτο. Γιατί αρχικά οι νομικέ υποχρεώσει μιλούσαν μόνο για υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή του κανονισμού. Αλλά καταλάβαμε ότι η εφαρμογή πραγματικά είναι ε, ένα σημαντικό τομέα. και αφορά και τομεί που δεν συνδέονται άμεσα με τον κανονισμό, αλλά που σίγουρα θα άξιζε τον κόπο να ασχοληθούμε εμεί με αυτού για του πολίτε τη Ευρώπη. Λίγα λόγια για το υπόβαθρο γιατί υποβάλαμε αυτή την ανακοίνωση. Γιατί όπως σας είπα η επιβολή είναι μία από τους, ένας από τους πυλώνες ε, του, της στρατηγικής για την κατανάλωση για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ε, 2007 στο 2013. Τέλος, επίση, ε, επίσης οι προκλήσεις που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε σχετίζονται με την εφαρμογή. Και τρίτον, η νομική υποχρέωση για την υποβολή εκθέσεων προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οπότε μας προέκυψε αυτό το πακέτο. Λίγα λόγια για το δίκτυο CPC που αναφέρατε ήδη, τα SWIFT που είναι πραγματικά ένα βαρχίδα των προϊόντων ε, και που επικεντρώνει τις πιο προφανείς δράσεις ως προς αυτό. Το δίκτυο τι είναι. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είμαστε στην διαφάνεια 3 ε, εκεί είμαστε. Όχι την προηγούμενη. Είναι λειτουργικό λοιπόν από τον Δεκέμβριο 2006 όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο κανονισμός ε, για, το, για τους κατραλωτές. Είναι ένα μέτρο που αφορά τις ε, αρχές, τις εθνικές αρχές που δίνει, τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο το, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως λέει πολύ καλά, είναι κοινή αρμοδιότητα αυτή για να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη τους ε, νόμους και η Κομισιόν υπάρχει για να δίνει το ε, πλαίσιο για τη λειτουργία του δικτύου αυτού. Το δίκτυο CPC τι κάνει, τι μπορούν να κάνουν αυτές οι αρχές για μας. Καταρχήν, μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Αυτό είναι το το κωδικό όνομα για τις ε, έρευνες. Αν δηλαδή θεωρήσουν ότι αρξίζει κάτι διερεύνηση σε μια άλλη χώρα, μπορούν να ξεκινήσουν αυτή τη διερεύνηση. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν εφαρμοστικά μέτρα. Αν το συλλογικό καλό διακυβεύεται των κατανοτών, τότε μπορούν να ζητήσουν στους συναδέλφους ε, των άλλων χωρών να, σταματήσουν την ε, παραβίαση με οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει στο δικό του εθνικό δίκαιο. Επίση, όταν σε, πρώιμο, σε πρώιμη φάση διακρίνουν κάποιο κίνδυνο, όχι άμεσο για κάποια άλλη χώρα, αλλά ε, δυνατότητα αντιγραφή ε, και που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τους κατανοητές άλλων χωρών μπορούν να ενημερώσουν η μία χώρα την άλλη και να δοθεί απαραίτητη υποστήριξη έτσι, η απαραίτητη βοήθεια το πεδίο εφαρμογή είναι περιορισμένο του δικτύου. Το δίκτυο και ο κανονισμός υπάρχουν για να προστατεύσουν το συλλογικό καταναλωτικό καλό και να ενισχύσουν τις οργανώσεις, ειδικά όταν πλήττεται ή πρόκειται να πληγεί το συμφέρον των καταναλωτών. Επόμενη διαφάνεια. Τι κάναμε. Σα είπα ότι το δίκτυο λειτουργεί από το 2006. Το 2007 ήταν η πρώτη, το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του. Ε, διαχειριστήκαμε 327, 327 αιτήματα, το 2008 392 αιτήματα, εκ των οποίων 100 ήταν προειδοποιήσει Φέτος που δεν είναι βέβαια τμήμα της έκθεσης, γιατί καλύπτονται μόνο τα δύο χρόνια λειτουργία στην έκθεση, φέτος ήδη έχουμε διαχειριστεί περίπου 300 αιτήματα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε στα ίδια επίπεδα μέχρι να τελειώσει και αυτό το έτος, στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλο κάνουμε. Γιατί εδώ μιλούμε για τη διαχείριση των ε, ε, περιπτώσεων. Είναι η καθημερινή δουλειά των αρχών. Αλλά θέλαμε να ε, έχουμε και κάτι παραπάνω που να είναι λίγο πιο προφανές και πιο αξιόλογο και που μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους. Το πρώτο λοιπόν, ήδη αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο, ήδη οργανώσαμε τρεις, ε, τρία συντονισμένα εγχειρήματα επιβολής που τα ονομάζουμε SWIPs. Αυτές είναι δράσεις όπου οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν το ίντερνετ, τις αγορές online, τις ιστοσελίδες, ελέγχουν κατά πόσο συμβαδίζουν με το νομικό πλαίσιο και αν χρειαστεί αναλαμβάνουν δράση. Επίσης, κάνουμε κάποια κοινά προγράμματα. Όταν οι διάφορες αρχές από τις ε, χώρες συνέρχονται, μπορούν να θέσουν ένα στόχο κοινό, ο οποίος συγχρηματοδοτείται και από το εθνικό και από τον κοινωτικό κορβανά. Και τρίτον, Η λειτουργία του δικτύου δίνει πραγματικά πολύ χρήσιμα δεδομένα για την χάραξη της πολιτικής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται και για τον πίνακα για τις αγορές των καταναλωτών. Αλλά χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά και ως δείκτες για να τονίσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στην ε, εφαρμογή της ιστορικής αγοράς. Αυτό κάνουμε. Και αυτό κάναμε. Έχουμε πάνω από 300 αρχές ε, επιβολής στην Ευρώπη. Έχουμε περίπου χίλιους, ε, ε, χίλια άτομα που ασχολούνται στην Ευρώπη. Οπότε πραγματικά είναι μεγάλο το δίκτυο και αντιπροσωπεύει, έχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Το πακέτο τώρα υιοθετήθηκε 2 Ιουλίου του 2009 και καλύπτει δύο πρωτοβουλίες. Μία είναι η ενημέρωση και η άλλη είναι η έκθεση ε, η διετής, ε, σύμφωνα με την οποία πρέπει κάθε δύο χρόνια να αξιολογούμε την λειτουργία του δικτύου. Η πρώτη είναι μια πρωτοβουλία γιατί είδαμε τόσα πολλά νέα στοιχεία, τα οποία δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογή της διετούς έκθεσης, οπότε ήταν, θα ήταν κρίμα να τα χάσουμε, γι' αυτό ε, αναφέρουμε αυτή την ανακοίνωση εδώ. Η ανακοίνωση τώρα. καθορίζει το υπόβαθρο, δηλαδή δίνει ορισμούς για την επιβολή, εφαρμογή του νόμου, καθορίζει ποιε είναι οι βασικές προκλήσεις και καθορίζει και τις, ε, τους τομείς δραστηριότητα. Τους τομείς προτεραιότητας, συγγνώμη, για δράση. Επίσης, καθορίζει πέντε τομείς προτεραιότητα. Θα σας τους αναφέρω βεβαίω. Και μια που είναι νέος ο κανονισμός αυτός, δεν θέλαμε να οδηγηθούμε σε καμία, σε καμία νέα νομική πρωτοβουλία. για να δούμε πώ μπορούμε. Δεν θέλαμε δηλαδή καινούργια πράγματα, θέλαμε να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε για να βελτιωθούν τα πράγματα. Οι πέντε τομεί προτεραιότητα είναι, χωρί καμία ιδιαίτερη αξιολογική σειρά, Καταρχήν, να ενισχύσουμε τα πλαίσια ε, συνεργασίας. Έχουμε δύο τέτοια πλαίσια. Το ένα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των ε, προϊόντων, το RAPEX, και το άλλο για προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, το δίκτυο CPC. Δεύτερο, δεύτερος τομέας, ενίσχυση της διαφάνειας της εποπτείας αγοράς και εφαρμογή των διαρευνήσεων. Από τους ε, ανθρώπους που ασχολούνται ε, με την εφαρμογή μας είπαν ότι το πιο χρήσιμο εργαλείο είναι η δημοσιότητα. Έχει δύο πλεονεκτήματα. Καταρχήν, μπορεί να προειδοποιήσει πιθανά ενδεχόμενα θύματα, καταναλωτές, μπορεί να, και μπορεί να το, τα ευαισθητοποιήσει. Και δεύτερον, μπορεί να βρει εταιρείε, επιχειρήσεις που θα ε, έμπαιναν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δραστηριότητε που δεν επιτρέπονται. Η δημοσίευση στέλνει αυτό το μήνυμα ότι υπάρχει ένα δίκτυο και μπορεί να ε, εποπτεύσει, οπότε καλύτερα να το σκεφτούν δύο φορές αν θέλουν όντως να δράσουν παράνομα. Ε, είναι πιο λειτουργικό το σύστημα αυτό για να μπορέσουμε να εργαστούμε ώστε να εκπονηθεί ένα κοινό, μια κοινή δέσμη κανόνων για τους καταναλωτές. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες βεβαίως, αλλά καμιά φορά υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή τους, στη μεταφορά στα κρατημέλη, οπότε ήταν, θεωρήσαμε απαραίτητο, όπως μας είπαν οι επιβολείς του νόμου στα διάφορα κράτη-μέλη, να καθορίσουμε κάποιους ορισμούς Χρησιμοποίησαμε τα sweeps γι' αυτό, έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και έχουμε και τις κοινέ δραστηριότητε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ο τέταρτος τομέας, ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς για να, στόχο, για να ε, επιτύχουμε τον στόχο αυτό που είναι η καλύτερη εφαρμογή. Έχουμε και το scoreboard των αγορών, πάνω στο οποίο θα εμφασίζουμε τις ε, αποφάσεις για το μέλλον. Δηλαδή θα έχουμε απόλυτα στατιστικά στοιχεία. Και επίσης, η Ευρώπη είναι μεγάλη και μεγαλώνει κι άλλο. Αλλά δεν είναι αρκετά μεγάλη. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις απειλές και τις προκλήσεις που προέρχονται απ' έξω. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητη η διεθνής ε, συνεργασία. για το μέλλον. Στην, ε, στον τομέα της προστασίας των αγαθών ισχύει, για το RAPEX δηλαδή, ισχύει με την Κίνα και τον Καναδά και στο CPC ε, ισχύει, διαπραγματευόμαστε μάλλον μια συμφωνία συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Αυτά λοιπόν είναι τα πορίσματα της ανακοίνωσης. Πάμε τώρα στην ε, έκθεση, τη διετή. Εδώ έχουμε μια σαφή νομική υποχρέωση για, υποβολή εκθέσεων ε, κάθε δύο χρόνια, δυνάμει του άρθρου 21. Αυτή η έκθεση συνδέει τις απόψεις των κρατών μελών και τις απόψεις της Κομισιόν για την εφαρμογή του CPC και του σχετικού κανονισμού και μια που πρέπει να καλύπτονται δύο χρόνια, καλύπτονται αυτή τη φορά το 2007 και το 2008. Σε αυτή την έκθεση, το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι το δίκτυο CPC ήδη δίνει αυτά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Είπα ήδη ότι έχουμε διαχειριστεί 700 περίπου ε, περιπτώσεις ε, στα πρώτα δύο χρόνια. Αλλά βλέπουμε ότι φυσικά δεν έχουμε φτάσει στο 100% των ε, δυνατοτήτων του δικτύου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και αυτά προσπαθούμε να λύσουμε. Βρήκαμε δύο βασικά, βασικές ελλείψεις. Ένα είναι τα επιχειρησιακά θέματα και το δεύτερο τα οριζόντια θέματα. Μιλούμε λοιπόν για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να είναι καλύτερη η εφαρμογή για να έχει καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των καταναλωτών. Και τέλος, ποια είναι τα επόμενα βήματά μας. Πώς θα προχωρήσουμε. Καταρχήν, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τις αρχές για να αντιμετωπιστούν τα επιχειρησιακά θέματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε την ε, επιβολή του νόμου πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική. Έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. εμείς ε, ως Κομισιόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τα κρατημέλη, γιατί τα κρατημέλη είναι αυτά που εφαρμόζουν. Οπότε χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ μας. Και δεύτερον, σίγουρα Χρειάζεται να είναι λειτουργικό το δίκτυο και ε, να λειτουργεί αποτελεσματικά. Και αυτό έχει να κάνει με πόρους. Οικονομικούς πόρους, ανθρώπινους πόρους και πολιτική δέσμευση. Αυτό είναι ο τομέας που θεωρούμε ότι ακόμη μπορούμε να βελτιώσουμε κατά πολύ τα πράγματα στην Ευρώπη. <coughs> Και το δίκτυο η λειτουργία του πιστεύουμε ότι μπορεί να ενισχυθεί χωρίς να χρειαστούν άλλα νομικά, άλλες νομικές δράσεις. Αυτό λοιπόν είναι το πακέτο, αυτά είναι τα δύο έγγραφα και ευχαρίστως να απαντήσω σε οτιδήποτε, σε όποιο ερώτημα σας ε, προκύψει. Anyway, thank you very much indeed. I thought it was uh, a very clear presentation. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ ξεκάθαρα μας τα είπατε και ενημερωτικά πολύ θα τα έγραφα. Οπότε τώρα συνάδελφοι, εσείς έχετε τώρα τη σκητάλη για παρατηρήσεις, σχόλια. Η κυρία Γκέμπχαρτ πρώτη έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Μούζης μετά. Οπότε έχει ανοίξει ο κατάλογος των αγορητών. Κρότσμαν. Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Άρα η Ευλίνγκη θα λάβει πρώτη το λόγο για να μας πει για τον εφαρμοστικό κανονισμό, κείμενο για το οποίο είναι υπεύθυνη για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την ε, πολύ <clears throat> ξεκάθαρη παρουσίαση των προβλημάτων που έχουν αναγνωρίσει Κάποιοι από τους συναδέλφους μου δεν ήταν, ε, δεν ήταν τότε στο κοινοβούλιο, οπότε θα σας θυμίσω μερικά πράγματα. Τότε πρόκειτο για τη διοικητική συνεργασία ή, εν πάση περιπτώσει, τη συνεργασία των ε, αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή του νόμου και, την, και τη λύση προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά των καταναλωτών. Σε αυτόν τον κανονισμό Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι, λίγο, είναι αρκετά γραφειοκρατικό, είναι αρκετά επαχθές και που δεν μας είχε αρέσει ούτε τότε όταν το αποφασίσαμε, αλλά τότε ήταν η μοναδική δυνατότητα που είχαμε για την συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Να έχουμε δηλαδή κάτι που να μπορεί να προχωρήσει. Και αυτό οφειλόταν στο εξή. Οι αρχέ των κρατών μελών, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου, είχαν τελείως διαφορετικούς τρόπους για να γίνει αυτό. Και πολλές φορές ήταν και η επιβολή επαφίετος σε διαφορετικές αρχές. Θυμάμαι πάρα πολλέ συζητήσεις μεταξύ Γερμανία και Ηνωμένου Βασιλείου, όπου εκεί υπήρχαν πραγματικά οι μεγαλύτερε ε, δυνατότητες για να ε, προχωρήσουν σε έναν κοινό δρόμο αυτές οι δύο χώρε Στη Γερμανία η νομική η τάξη ήταν τελείως διαφορετική από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλούσαμε πάντα για δημόσιες αρχές. Οι Βρετανοί δεν μπορούσαν να φανταστούν λοιπόν συνεργασία με έναν οργανισμό ή μη, μια μη κυβερνητική οργάνωση που ήταν το, η παράδοση στη Γερμανία και αυτά ήταν τα βασικά προβλήματα που έπρεπε τότε να διαχειριστούμε. Γι' αυτό είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα έτσι ώστε να υπάρχει κάτι έστω ώστε να διευκολύνει την συνεργασία. Γι' αυτό δεν περίμενα ότι μετά από μια έκθεση και δύο χρόνια θα είχαμε την αναθεώρηση ας πούμε της νομοθεσίας γιατί ε, είναι σαφές ότι εδώ είναι, υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Πρέπει να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Ότι δηλαδή είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ τους. Και είναι σαφές ε, μέσω της παρουσίασής σας ότι στον τομέα της λειτουργίας ακόμη υπάρχουν ε, πολλές δυνατότητες για βελτίωση. Και γι' αυτό είναι καλό που έχουμε αυτές τις εκθέσεις, έτσι ώστε ως Κοινοβούλιο να έχουμε τη δυνατότητα να τις ε, μελετήσουμε προσεκτικά, να δούμε πού είναι τα προβλήματα και ένα από τα ερωτήματα που έχω προς εσάς είναι αυτό ακριβώς. Μας είπατε έτσι πολύ ωραία ότι υπάρχουν κάποια λειτουργικά προβλήματα ή δυνατότητες βελτίωση. Ποια είναι όμως αυτά τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Και επίσης, ποιες είναι οι δυνατότητες επίλυσης τους, εκτός δηλαδή όσων εκτός των ε, οικονομικών θεμάτων και των θεμάτων ανθρωπίνων πόρων στα κρατημέλη, που ούτως ή άλλως παίζουν ρόλο. Και με την κρίση τώρα που περνούμε, φαντάζομαι ότι το οικονομικό θα είναι ένα από τα βασικά προβλήματα για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θα ήθελα εγώ να θέσω. Και δεύτερον, Μα δώσατε κάποια νούμερα για το 2007 και 2008 και για το 2009 για τα αιτήματα που υπευλήθησαν αλλά δεν μας είπατε τίποτα για το κατά πόσο ήταν επιτυχή όλα αυτά ή τέλο πάντων ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των ε, ερωτημάτων και εγώ θα ήθελα πραγματικά να μάθω, θα με ενδιέφερε να μου πείτε το 2007 είχατε 327 ε, ερωτήματα. Πού ήταν καλύτερα η συνεργασία, πού δεν πήγε καλά και από αυτά τα 327 πόσα τελικά κατέληξαν με θετικό αποτέλεσμα. Και πόσα δεν κατέληξαν σε τίποτα. Και σε αυτά που δεν κατέληξαν σε τίποτα, γιατί δεν κατέληξαν σε θετικό αποτέλεσμα και γιατί δεν εξευρέθη η λύση. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πραγματικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μας δώσετε δύο-τρεις πληροφορίες. Και τρίτον και τελευταίο, για τα λειτουργικά ήδη τα είπα, θα μπορούσατε να μας πείτε, εκτός από τα συστήματα με το RAPEX, το CPC, το Scoreboard, τα SWIPS, εσείς από τη δική σας ε, γνώση, από τις έρευνες που κάνατε, από την εμπειρία σας, τι άλλο θεωρείτε ότι χρειάζεται. Και αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ θα μπορούσε να δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν ε, τέτοιοι μηχανισμοί ε, συλλογικοί, ευρωπαϊκοί για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σωστή συνεργασία και σε όφελος προς τους καταναλωτές. Αυτά από ένα πρόεδρο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε για αυτές τις ερωτήσεις. Θα ακούσουμε και κάποιες ακόμη και με βεβαίως ότι η, κυρία, ότι η Επιτροπή τη σημειώνει. κυρία Σάντε Ja, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ήταν συναρπαστικά όσο ακούσαμε. Όμως νομίζω ότι εγείρουν, εγείρει πολλά ζητήματα η παρουσίαση σας. Όπως αυτές οι 700 υποθέσεις που εξετάσατε, τι περιπτώσεις είναι. Ποια είναι τα ποσά που εμπλέκονται εδώ και πώ επιλύθηκαν οι διαφορέ χάρη στη συνεργασία μεταξύ των κρατών Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να έχουμε εδώ κάποιε λεπτομέρειε, διότι στην Δανία σημειώνω ότι εισαγάγαμε ένα τέτοιο σύστημα και σε πολλέ περιπτώσει χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να λειτουργήσει όλη η διαδικασία. Οι ιστότοποι των αεροπορικών εταιριών λόγου χάρη δεν σέβονταν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έπρεπε λοιπόν να παρέμβουμε και να απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Αλλά υπήρξε τεράστια χρονική καθυστέρηση. Πέρασαν πάρα πολλοί μήνες μέχρι να επιληθεί οριστικά το ζήτημα. Εσείς λοιπόν τι χρονικό πλαίσιο προβλέπετε Μήπω αυτό είναι πραγματικά το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Για τι περιπτώσεις λοιπόν μιλάμε, αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Και έπειτα να συμφωνήσω μαζί σας ότι εάν θέλουμε το σύστημα να λειτουργήσει θα πρέπει να δεσμεύσουμε περισσότερα κονδύλια και με τέτοια να πρικοδοτήσουμε τι αρχέ επίβλεψη τη αγορά των 100 μελών. Ε, είναι απαραίτητο αυτό για την υλοποίηση μια πολιτική. Πριν από λίγε εβδομάδε, άλλωστε, είπαμε και ακούσαμε την Επιτροπή να λέει ότι για την υλοποίηση των μέτρων επίβλεψη τη αγορά, μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να αποδεσμεύσουν περισσότερα κονδύλια για αυτού του σκοπού. Δύο λοιπόν αυξάνουν τα ποσά για να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα επαγρύπνηση τη αγορά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολήσει. Η επίβλεψη της αγοράς είναι καθοριστική σημασία αν θέλουμε να έχουμε επιβολή. Επιτυχή. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω. Όλες οι οδηγίες μας και όλοι οι κανονισμοί δεν ισχύουν, δεν αξίζουν τίποτα δεν υπάρχει ένα σύστημα υποπτίας. Να, να δούμε δηλαδή τι γίνεται, τι κάνει κανείς και πώς μπορεί να αποφύγει την γραφειοκρατία η παρακολούθηση όντως ε, μπορούμε να την βελτιώσουμε. Ε, μπορούμε να τη βάλουμε στον πυρήνα της συζήτησης, ε, να δούμε ποια είναι η καλύτερη πρακτική ίσως από κάποιο κράτος μέλος, να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία όλων. Η στοχευμένη, προ, η στοχευμένη έλεγχη στα σημεία πρόσβαση επίσης είναι θέμα. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε ας πούμε Ρότερνταμ, Αμβούργο, Γένοβα. Ε, πρόσβαση από χώρε εκτό τη Ένωση. Αν δεν υπάρξει κανένα ε, έλεγχο εκεί, που δεν γίνεται γιατί είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσει. είναι πάρα πολύ δύσκολο εντό των χωρών να γίνουν οι έλεγχοι και να ανακαλυφθούν ότι όποιες παράνομες δραστηριότητε ε, γίνονται. Και το θέμα είναι πώς θα ενισχύσουμε τους ελέγχους στα κράτη και πώς μπορούμε, αν υπάρχουν όντως προβλήματα στα σημεία εισόδου, να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Να έχουμε, ας πούμε, κάποιους ελέγχους σε κάποια λιμάνια και τα ε, και τα εμπορεύματα να περνούν από, από ε, λιμάνια τα οποία δεν ε, την χάνουν επισχυρών ελέγχων και να αποφεύγουν όλα τα υπόλοιπα λιμάνια τα, στα οποία γίνονται σημαντικοί έλεγχοι. Οι εισαγωγείς πάντα μπορούν να το κάνουν αυτό για να ξεφύγουν. Οπότε πρέπει να το, να το δούμε. Είναι σαφές ότι τα λιμάνια πρέπει να κάνουν εντατικούς ελέγχους. Γιατί εκεί υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Βεβαίω, αυτό έχει σχέση και με το κόστος. Έχει όμως σχέση και με την αποτελεσματικότητα. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η έλεγχη, τόσο πιο αποτελεσματικά θα είναι και, τα, και η αντίδραση των λιμένων και τόσο πιο πολλά χρήματα θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον συναδέλφους. Είναι πολύ σαφής η παρουσίαση της Κομισιόν για το δίκτυο των καταναλωτών. Όντως είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τώρα πόσο επιτυχές ήταν το δίκτυο αυτό στα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό να ε, υιοθετήσουμε μια σειρά μέτρων ε, σε ένα πιο γενικό πλαίσιο και έτσι να, προ, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ε, κατά τη και την ε, ευρωπαϊκή αγορά έναντι των παγκοσμίων αγορών. Νομίζω η κυρία Κούνεβα το είχε πει, ειδικά σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς και τους Κινέζους για το ράπεξ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Και δεύτερον, όταν θα συζητήσουμε την έκθεση της κυρίας Χέντ, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το Consumer Market Scoreboard και πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα προβλήματα και να απαντήσουμε και στα ερωτήματα που τίθενται. Και χωρίς να θέλω να επανέλθω σε αυτές τους πέντε τομείς προτεραιότητας που έθιξε η Κομισιόν, ερώτημα, η Κομισιόν τι μας προτείνει για την περαιτέρω ανάπτυξη του scoreboard, αυτή την εργασία του Κοινοβουλίου πώς μπορούμε να την ε, ενσωματώσουμε καλύτερα σε, αυτή την, ε, σε αυτό το δίκτυο εφαρμογής του καταναλωτικού κεκτημένου. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Σας πω και εγώ μια-δυο παρατηρήσεις και κατόπιν να απαντήσει ό,τι ερωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως έχουμε και ακόμα γύρω τρόπες. θέλαμε να συνδυάσουμε και το άλλο θέμα τη κυρία της κυρίας Head ως αυτό το scoreboard διότι είναι ελένδετα συνδεδεμένο όμως σήμερα είναι άρρωστη και έτσι δεν μπορούμε. Κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση τώρα που κοιτάω την ανάλυση της έκθεσης είναι ότι ήταν κάπως εμβαλωματικές οι παρατηρήσεις που έγιναν από τα κράτη-μέλη ούτε το θέμα συνδέθηκε με το μέγεθος των κρατών μελών. Αυτή η αιτήση της αμοιβίας για τα κρατή-μέλη, η Δανία υπέβαλε 14 το 2008, η Ιταλία 2, η Δεγαλία 16. Επομένως ε, είναι, υπάρχει ανισότητα στην αντιμετώπιση να θέμα τεχνολογία ίσως. Είπατε ότι είναι θέμα μεγαλύτερων επενδύσεων. Άρα θα πρέπει να πιστούν τα κρατημένα να επενδύσουν περισσότερο. Επίσης μας τονίσατε ότι αυτή η υπόθεση αφορά περισσότερο όχι μόνο περιπτώσεις, αλλά συλλογικά θέματα. Έχουν υποβληθεί και κάποιες ε, αναφορές από κάποια φυσικά πρόσωπα, άρα ίσως είναι και διασυνοριακές ε, υποθέσεις αυτές. Για να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές επί των διαφορετικών συστήματων δικαίου, διαφορετικών κρατών. Επίσης για κάποιες ομαδικές ε, αγωγές ε, είχε κάποιες προτάσεις η Κομισιόν, έτσι παρεκτάθηκε το πεδίο Έχουμε κάνει τη σχετική έκθεση με αυτές τις αγωγές. Μήπως μπορούμε να μας πείτε δύο λόγια πώς θα μπορούσε αυτό το σύστημα να λειτουργήσει. Αυτές οι ομαδικές αγωγές των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ, λέει πρόσωπο της Επιτροπής. Μερικές ερωτήσεις αφορούν το ίδιο θέμα. Μερικές όχι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και όπως είπατε, εάν υπάρχει χρόνος για δεύτερο γύρο τραπέζι, θα δούμε. Επομένως, για μένα το πιο σημαντικό θέμα εδώ είναι το τι θέλουμε να δώσουμε στον πολίτη. Γιατί χρειάζεται αυτό το δίκτυο, γιατί χρειάζεται η εφαρμογή, επιβολή του νόμου, γιατί θα πρέπει να κατοχυρωθούν εδώ τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτό δεν αμφισβητείται ότι έχουν δικαιώματα οι καταναλωτές. Θεωρείται καλό. Όμως, ταυτόχρονα, έχω την αίσθηση ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των καταναλωτών δεν, είναι, δεν έχει την ίδια προτεραιότητα από πλευρά κυβερνήσεων όπως άλλα θέματα. Και γι' αυτό μιλήσαμε για πόρους, για χρόνο που χρειάζεται ώστε να γίνει επιβολή νόμου, για μία σειρά ζητημάτων που επιδιώκει κάθε χώρα, τις δικές της προτεραιότητες. Τι γίνεται όμως, είναι πραγματικά προτεραιότητα ε, ε, για τις αρχές κάποιες χώρες τόσο ώστε να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Σε οποιαδήποτε χώρα. Είναι προτεραιότητα για ένα κράτος ή όχι. Τότε το παίρνουν στα σοβαρά και κάνουν τα απαραίτητα βήματα. Ε, γι' αυτό είπαμε ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν καθορίζει το πόσες φορές έχει ζητηθεί αρρωγή, έχουν προσφύγει στην ε, αρχή αυτή οι χώρα Εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να επισημάνουμε. Είναι και θέματα πολιτικής προτεραιότητας κυβέρνησης. Πάντως, κοινό αγώνα κάνουμε. Είστε κι εσείς στόχο τον ίδιο με εμάς. Τώρα. να δούμε τι ε, λύσεις μπορεί να υπάρξουν για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Και ποια είναι αυτά. Είπαμε, είναι ζήτημα ανθρώπινων πόρων και χρηματικών πόρων, τα οποία ζητήματα αυτά είναι αλληλένδετα. Επίσης, είπαμε ότι δεν εμπλέκονται όλες οι συναρμόδιες αρχές για την προσβασιμότητα στο σύστημα είναι intranet, δηλαδή θα πρέπει κανείς να έχει έναν υπολογιστή με καλώδιο και να συνδεθεί με το καλώδιο. Και μετά κάθεται κανείς στο κομπιούτερ και μπορεί να επικοινωνήσει σε κάποια γλώσσα με τους άλλους αδέλφους του, αλλού στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνεπάρχουν αλλιώ. Είναι δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τους συναδέλφους του. Άλλα σημαντικά θέματα, νομίζω ότι αναφέρθηκε από την κυρία Γκέμπχαρτ, ότι τότε προσπαθούσαμε μαντεύοντας να βρούμε τι χρειάζεται, τι, τι μορφή έλαβαν τα πράγματα. Προσπαθούσαμε να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις. Τι συνέργεια θα διαμορφωθεί. Τώρα πέρασαν τόσα χρόνια. Οπότε έχουμε την εμπειρία και έτσι μπορούμε να τροποποιήσουμε τους εφαρμοστικές διατάξεις. Να είναι πιο στοχοθετημένες οι κινήσεις μας. ψάχνει κανείς την ε, βάση δεδομένων ε, η μία αρχή να μπορεί να βρει την άλλη η Επιτροπή επίσης μέσα από αυτές τις βάσεις δεδομένων τώρα για το τι κάνουμε τι, τι, τι υποθέσεις μας απασχολούν δεν μπορώ να σας πω γιατί ούτε από πλευρά Κομισιόν δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο σύστημα έτσι. Δεν μπορώ να κοιτάξω. Εντάξει, αυτό τα ξέρουν οι διοικητικές αρχές, οι αρχές της επιβολής, της εφαρμογής του νόμου. Τρία διαφορετικά sweep συντρέχουν. Ένα σε κάποιο website που πουλούσε αεροπορικαστήρια, το άλλο ηλεκτρονικά. Και η τρίτη περίπτωση αφορούσε κάποια ιονή λογισμικά για κινητή τηλεφωνία. Οπότε, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τομείς που εμπλέκονται εδώ. Από πλευρά στατιστική μπορούμε να πούμε ότι η οδηγία ε, όπου σημειώνει πιο πολλές παραδιάσεις, είναι η οδηγία η σχετική με την παραβίαση των κανόνων άσκησης του εμπορίου. Άρα, πάντα από πλευρά στατιστικής μπορώ να σας πω ενδεικτικά ότι κατά μέσο όρο οι ημέρες που ε, είναι μέρε που ασχολούμεθα με κάποια συγκεκριμένα αιτήματα, είναι περίπου 150 μέρε. Δεν ξέρω αν αυτό σα φαίνεται υπερβολικά λίγο, υπερβολικά πολύ. Κρίνετε εσείς. Σε πέντε λεπτά, αν θέλω, αλλάζω το περιεχόμενο του website. Όμως, εάν είμαι αρχή, χρειάζομαι έντελμα. Πρέπει να πάω σε δικαστή. Μπορεί ο εγκαλούμενος, ο κατηγορούμενος να ασκήσει έφεση και λοιπά και για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έχουμε τα μέσα που χρειάζονται. Τα νομικά μέσα και εργαλεία, ούτως ώστε μπορούμε ταχύως να επέμβουμε. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις διαδικαστικές προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. και αν ε, αυστηρά τηρήσουμε τις σχετικές προθεσμίες μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει δουλειά. Να πούμε σε ένα επιχειρησιακό λειτουργικό θέμα. Ότι θα πρέπει επομένω έτσι να ε, συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου. Επίση, υπάρχουν κάποια εργαστήρια με ε, συγκεκριμένα θέματα όπως ας πούμε για το εφαρμοστέο δίκαιο, τι θα πρέπει να ισχύει κάθε φορά που έχουμε κάποια παραβίαση. Υπάρχει ένα άλλο εργαστήριο το οποίο φέρει αφορά τι κυρώσει. Ε, Επίση, μισή μέρα ασχοληθήκαμε για το κατά πόσο πρέπει κανεί να κατονομάζει του υπόπτου, του φερόμενου ω υπόπτου, μέχρι ότου ε, ληφθεί κάποια τελεσίδια από δικαστήριο. Όλα αυτά τα ζητήματα επομένω ε, απασχολούν τις ε, αρχές επιβολής του νόμου στην Ευρώπη. Και εγώ όλα αυτά τα συζητούμε με ανοιχτό τρόπο. Τι μπορούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, η επιβολή του νόμου αποδίδει ή όχι. Από 700 υποθέσεις που σας προανέφερα, λιγότερο από το 10% των υποθέσεων ε, κρυμούν για περίοδο μεγαλύτερη του έτους. Από τις 700 όμως είχαμε 60 που σας ανέφερα που έμειναν χθες πάνω από μία χρονιά. Ίσως τώρα κρεμούν ενώπιον δικαστηρίου, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι αρχές επιβολής του νόμου. Τέλος πάντων δεν, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Στις 2 Δεκεμβρίου θα έχουμε ένα εργαστήριο για το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Να άρουμε τα εμπόδια, κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό το οποίο είπατε. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει βοηθεία τη αγορά ή των αγορών. Νομίζω ότι οι αρχέ επιβολή του νόμου κάνουν καλή δουλειά. Νομίζω και για το CPC και για την ασφάλεια των προϊόντων είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία έχουμε και δουλεύουμε. Επομένω, θα πρέπει όλοι, σε όλα τα κατημήλια, να ασχοληθούν όσο γίνεται περισσότερο με την εκδοχή του νόμου, να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότερε δραστηριότητε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μοιραστούν τι ε, θετικέ του εμπειρίε με του άλλου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο αποτελεσματικό μέσο πολιτική που έχουμε σήμερα. Το να μοιράζεται κανεί την εμπειρία του με του συναδέλφου, α πούμε για τα προϊόντα χαμηλή ποιότητα να βρεθεί ποιος είναι ο κρίκος στην αλυσίδα. Γιατί άμα το βρουν αυτό οι παρανομούντες, τότε θα ρίξουν και όλα τα κακά προϊόντα και θα πλημμυρίσει η αγορά με αυτά τα κακά προϊόντα. Άρα έτσι θα πρέπει να μοιραζόμαστε τις τέτοιες εμπειρίες, τη γνώση, πληροφορία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Χρηματοδότηση οικονομική υποστήριξη για την συγκρότηση κάποιων ε, εργαστηρίων, κινητών που να μπορούν να πάνε όπου χρειάζεται. Και σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή του νόμου είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Αν θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό και το οποίο δεν ισχύει πάντα, γιατί έχουμε κάποιες περιπτώσεις που τις περισσότερες φορές θεωρούν ότι είναι θέματα αστικού δικαίου και όχι ποινικού. Οπότε και οι λιμενικές αρχές και οι συνοριακές αρχές δεν εισακούονται όπως σε άλλου είδους ε, παραδείας του νόμου. Γιατί τώρα έχουμε τόσο διαφορετικά στοιχεία από χώρα σε χώρα. Γιατί δεν σχετίζεται το αποτέλεσμα με το μέγεθο της χώρας είπε ο κύριος Χάρμπορ. Όχι σε αυτόν τον το πόσο σοβαρά παίρνει το ρόλο της η διοικητική αρχή, η αρχή επιβολής του νόμου. Πόσο προσωπικά το παίρνει ο επικεφαλής κάθε φορά κάποιες υπηρεσίες, κάποιες διεύθυνσεις. Αν το θεωρεί θέμα προτεραιότητας. Γιατί. Ο καθένας μπορεί να πει δεν συνεργάζομαι. Δεν με νοιάζει για τους άλλους να συνεργαστώ. Θέλω να προστατεύσω μόνο τους δικούς μου. Το οποίο δεν είναι και τόσο παράλογο, ιδίω στο πλαίσιο της σημερινή οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά τώρα αυτές τις ομαδικές αγωγές, αποζημίως και το πόσο είναι ένα καλό μέσο ή όχι, είπαμε ότι θα πρέπει να δουν οι φυσικές αρμοδιότητες στις αρχές επιβολής, CPC, για να μπορούν να ασκήσουν την ομαδική αγωγή κατά μιας εταιρεία ή μήνυση για λογαριασμό των καταναλωτών. εστω όμω οι πόροι. Και τι θα γίνει με την αποζημίωση. Θα πάει στα θύματα θα πρέπει να πάει σε έναν κουμπαρά τη χώρα Και ποια χώρα. Όλα αυτά τα ερωτήματα επομένω αναδύονται. Βλέπετε πώς μπορεί για το πιο απλό πράγμα να μπερδευτεί. Τελευταία τώρα. Τελευταία ερώτηση που δεν την κάλυψαν ήταν το σκόρμπορντ. Αλλά όπως είπατε προηγουμένω, προβλεπόταν να συζητηθεί σήμερα. Αλλά θα το ξανασυζητήσει η Επιτροπή σας εν ευθέτω χρόνο. Άρα Θα έρθει κάποιο συνάδελφο που ασχολείται με αυτό και θα σα απαντήσει. Σα ευχαριστούμε για αυτέ τι διεξοδικότατε απαντήσει σα. Νομίζω ότι η Εύλην θέλει να επανέλθει και ίσω χρειαστεί να ξανά απαντήσετε. Ω επικεφαλή εισηγήτρια έχετε το δικαίωμα να δευτερολογήσετε, κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επιμείνω. Τα ερωτήματα απαντήθηκαν πολύ καλά, πιστεύω. Δεν ε, έχω να κάνω κανένα σχόλιο από αυτόν. Αλλά μια σκέψη έτσι μου ήρθε, που ήθελα να την αναφέρω. Για τα κράτη-μέλη και την επιβολή μέσω διαφορετικών πρακτικών και μέσω διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων και γενικώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών δεν είναι η ανώτατη αξία για όλα τα κρατημέλη όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι το συμπέρασμα όλων αυτών που είπατε. Και η δική μου πρόταση πρόεδρε θα ήταν να κάνουμε μια προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και να δούμε τι έχουν κάνει τα κρατημέλη. Αυτή θα ήταν ίσως μια δυνατότητα που έχουμε εμείς ως Κοινοβουλίο, έτσι ώστε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη και να αναγκαστούν, ας πούμε, να το σκεφτούν, κατά πόσο δηλαδή αυτόν τον ε, κανονισμό τον οποίο συν, ε, υπέγραψαν και συνδιατύπωσαν, αν τον έχουν εφαρμόσει όπως πρέπει. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, Πρόεδρε. Έτσι μια σκέψη που έκανα ήθελα να σας αναφέρω. Πολύ καλή ιδέα. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να συνεισφέρουν. Βέβαια, αναρωτιέμαι πόσοι από εκείνου γνωρίζουν τι δυνατότητε που προσφέρονται εδώ. Να ασχοληθούμε με περιπτώσει που θα του έχουν θέσει από την εκλογική του περιφέρεια. Να λοιπόν κάτι που μπορούμε να προβλέψουμε στο στρατηγικό μα προγραμματισμό για το 2010. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σα ευχαριστούμε. Ήταν εντελεχής η παρουσίασή σα. Θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε και την κυρία Χέντ που δεν ήταν εδώ. Και θα επηρεαστούν σίγουρα πολλέ από τι δικέ μα εργασίε από τα δικά σα στοιχεία. Συνάδελφοι τώρα, πρέπει να περάσουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για απόψε, πριν την συνάντηση των συντονιστών στις 5.30. Αυτό θα είναι η έκθεση για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση των εφαντουργικών προϊόντων. Εδώ η φέλτη κάθε Προέδρου είναι να λείπει ο εισηγητή από την αίθουσα. Ο κύριο Μάντερ αυτή τη στιγμή έχει εξαφανιστεί. Όμως θα φροντίσουμε να του στείλουμε ένα γραπτό μήνυμα για να εμφανιστεί. Έχουμε ίσως τους και όδης εισηγητές. Εάν μπορείτε λοιπόν να περιμένετε μαζί μας, η Σάλντερ Μόζε είναι εδώ. Ίσως να ακούσουμε πρώτα τους σκεώδεις, θα ήταν κάπως ε, ασυνήθιστο βέβαια. Και ας δώσουμε ένα λεπτό στον κύριο Μάντερς. Ελπίζω να έχει πάει στη σωστή αίθουσα. <laughs>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 Right, the missing rapporteur arrived. Έφτασε ο αγνώμενος εισηγητής. Ευτυχώς εγκαίρος. Έχετε αργήσει τρία λεπτά στις πέντε προβλέπονταν το θέμα σας. Αυτό το ρολόι πάει λίγο πίσω. Όταν ε, μπήκατε κοιτάξαμε το απέναντι ρολόι. Κυρίε και κύριοι, με χαρά μου υποδέχομαι τον κύριο Μάντερ και ανοίγω τη συζήτηση για την ονομασία των κλωστοϊφαντολογικών προϊόντων και τη συναφή επισήμανση. Έχουμε μισή ώρα το πολύ για αυτό το θέμα, νομίζω. Αλλά επειδή δεν είστε διαθέσιμο την επόμενη εβδομάδα και θέλουμε να συνεχίσουμε την εξέταση του θέματο, θα πρέπει τώρα να συζητήσουμε. Η κυρία Σαλτεμόζα είναι εδώ για το ΕΛΚ. Ε, νομίζω η κυρία Ρούλε, η ακούραστη κυρία Ρούλε που έχει αναλάβει για όλα τα ντοσιά εδώ την παρέμβασή της, η κυρία Σβένσον, η κυρία Σαρντίνη. Νομίζω έχουμε την κυρία Χουάλντε από την ε, Επιτροπή. Κύριε Μάντερς, λοιπόν, με χαρά σας δίνουμε το λόγο για να μας ενημερώσετε που έχουμε φτάσει για αυτό το σημαντικό, με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Είχαμε μια ιδιαίτερη επικοδομητική συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές. Ο αριθμός των εισηγητών διωγγώνεται συνεχώς. Ευχάριστο αυτό. Επειδή υπήρξαν πολλές ερωτήσεις, για το τι θέλουν οι σκιώδει για την επισήμανση. Το συζητήσαμε σε εκείνη τη συνάντηση, όλο και περισσότερε απαιτήσει προβλήθηκαν. όλο και περισσότερε πληροφορίε ζητήθηκαν από ό,τι αρχικά νομίζαμε. Θεωρήσαμε λοιπόν συνετό να έχουμε πληροφόρηση από εμπειρογνώμονε για το τι είναι εφικτό, τι είναι επιθυμητό, τι είναι καλό για του καταναλωτέ και ούτω καθεξή. Για αυτό το σκοπό ζητήσαμε να εκπονηθεί μελέτη η οποία θα περατωθεί στις αρχές του Ιανουαρίου για το πώς να καλύψουμε την ε, ετικετοθεσία. Θέλουμε πανευρωπαϊκή ετικετοθεσία. Θέλουμε ετικετοθεσία βάσει της ΣΕΝ, της του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης. Θέλουμε εικονογράμματα. Και ένα άλλο ζήτημα που θα μας απασχολήσει και θα προκαλέσει πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τριγμούς είναι το αν είναι εφικτό και επιθυμητό να έχουμε και επισήμανση για το μέγεθος στα ρούχα και ενοποιημένο σύστημα μεγεθών. Γιατί ξέρουμε όταν αγοράζουμε ρούχα από τη μια χώρα στην άλλη ότι πολλές φορές τα μεγέθη διαφέρουν. Και επειδή υπάρχουν περισσότερε διασυνοριακέ πωλήσει πλέον από το παρελθόν, θέλουμε και εδώ να υπάρχει σαφήνεια για τι χημικέ ουσίε επίση. Και για τι απαιτήσει υγεία και ασφάλεια. Τι κάνουμε με αυτό. Σε μία ενιαία γλώσσα ή με εικονογράμματα. Για τα βιοκτώνα προϊόντα. Θα συζητηθεί αυτό σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τι θέλουμε. Τι είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο καταναλωτής ποια προϊόντα, ποια χημικά προϊόντα επηρεάζουν την ένδυση, τα ενδύματα, ποια είναι τα, ε, ποιες είναι οι παρενέργειες για το σώμα όταν φορούμε τέτοια προϊόντα, τέτοια ενδύματα. Οι εισηγητέ θεωρούν ότι είναι συνετό να γνωρίζουν περισσότερο και για αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε σε μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά θα έπρεπε να έχουμε πολύ γλωσσή επισήμαση. Είδαμε το παράδειγμα των μεγεθών ή αρκεί να αναφέρουμε το τεχνικό, την τεχνική ονομασία του υφάσματος της Ίνας η οικολογική επισήμανση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσε πολλέ απαιτήσεις για τους καταναλωτέ και εμεί τι θέλουμε, τι θέλουμε να έχουμε, οικολογική επισήμανση. Ε, η χώρα προέλευση. Πολλά είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα το δούμε λοιπόν στις αρχές του Ιανουαρίου το το θέμα αυτό και ελπίζουμε ότι στην Ολομέλεια του Μαρτίου, τη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου, θα είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη. Ε, ακόμη, η συνάδελφος Κόμη έχει προσφερθεί να ερευνήσει το θέμα επιτοπίως. Όχι με επίσημη επίσκεψη της Επιτροπής ΙΜΚΟ, αλλά έχουμε ακόμη κάποια κονδύλια στον προπολογισμό μας για να οργανώσουμε επισκέψεις άτυπες Ευχαριστούμε και για την πρόσκλησή σας και για τη διοργάνωση και το πρόγραμμα που προβλέψατε. Από το mail βέβαια προέκυψε μια παρανόηση για το ποιο θα επικοινωνήσει με ποιον. Όχι, είναι μια ιδέα πρωτοβουλία επίσκεψη στι κλωστουριφαντουργικέ βιομηχανίε, στου σχεδιαστέ, στου designers και θα δούμε και τι άλλο. Πάντω, ήδη υπάρχουν οκτώ μέλη που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και θέλουν να έρθουν μαζί μα. Νομίζω λοιπόν θα ήταν καλό να μελετήσουμε τα κλωστοϊφαντουργικά στην Βόρεια Ιταλία. Ε, ίσως ο καιρός δεν είναι τόσο ευχάριστο όσο το καλοκαίρι, αλλά εδώ μας ενδιαφέρουν τα υφάσματα. Δύο μέρες δεν είναι και τόσο κουραστικό. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η μελέτη όλων αυτών των ζητημάτων, όλου αυτού του θέματος, με οδηγεί στο να σας ενημερώσω σε ένα πρόγραμμα που ε, στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο ονομάζεται bridge, δηλαδή η οικοδόμηση των ραδιοσυχνοτήτων σε ένα διεθνές περιβάλλον, κάτι που αυτή τη στιγμή ασχολείται ειδικό με την ένδυση. Μπορεί δηλαδή κανείς να παρακολουθήσει την πορεία ενός προϊόντος από τη χώρα προέλευσης μέχρι το σημείο πώλησης, αλλά να συμπεριλάβει και πολλές πληροφορίες εντωμεταξύ στις ετικέτες. Όλα αυτά βασίζονται στις ραβδοτές ετικέτες, όπου λογικά συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες. Και ίσω κάτι από όλα αυτά να το αξιοποιήσουμε για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, αντί να γράψουμε τόσα πολλά πράγματα σε μία ετικέτα. Έτσι, ε, ε, κάθε καταναλωτής μπορεί να δει και να, καταλά... να προσέξει αμέσω τι είναι σημαντικό για αυτόν. Την ε, οικολογική ετικέτα, τη χώρα προέλευση και το καθεξή. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υπήρξε πρόταση τη Επιτροπή και νομίζω ότι σύντομα θα το συμφωνήσουμε για την εισαγωγή νέων ινών και την πιστοποίησή τους. Νομίζω ότι ως πολιτικοί θυνάντες θα πρέπει να αναλάβουμε την ευκαιρία αυτή, να βελτιώσουμε τη θέση των καταναλωτών και την εσωτερική αγορά να την καταστήσουμε καλύτερη για το μέλλον. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ίσως με τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, εάν μπορούμε. Θέλω να δείξουμε στους συνεργάτους μας, αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε για μια ενιαία Ευρώπη, ότι αυτό ακριβώς κάνουμε. Προ στιγμήν αυτή είναι η θέση στην οποία βρισκόμαστε και με τα χαράς να ακούσω τα σχόλια, προσθήκες προτροπέ, προτάσει των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάντερς. Ήταν ε, πραγματικά πολύτιμη παρουσία σα τελικά. Στην τελευταία σα πρόταση αναφέρατε και την πρόταση τη Επιτροπή, Καλό αυτό. Αλλά ήταν πολύ εφάνταστη όλη σα τοποθέτηση. Οπότε νομίζω ότι και εσεί και οι σκιώδει εισηγητέ θα πρέπει να καθορίσετε μια κοινή προσέγγιση. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν ταυτόχρονα ή απλώ να ασχοληθείτε με την πρόταση που έχουμε επιτάπητο και να φροντίσετε να προχωρήσει. Είναι δική σα η απόφαση. σω το κείμενο για του παρασκευαστέ να μα οδηγήσει να του ρωτήσουμε και εκείνοι τι θέλουν. Διότι φαντάζομαι ότι εκείνοι αυτό που θέλουν είναι να εγκριθεί η πρόταση όσο το δυνατόν συντομότερα. Αλλά εσεί αποφασίζετε. Πολύ διασκεδαστική όμως παρέμβασή σα Ευχαριστώ. Και πολύ σοβαρή ελπίζω. Ναι, ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πραγματικά. Κυρία Κόμη. Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδες εισηγητές, με τους οποίους συνεργαζόμαστε κατά τρόπο άριστο. Οι προτάσεις που μόλις ανέφερε ο εισηγητής, ο κ. Μάντερς, είναι πολύ άριθμες. Είναι υψηλού επίπεδου και εξίσου σημαντικές. Σημαντικές διότι ακριβώς ο κλωστοϊφαντουργικός τομέας αφορά με πολλούς τρόπους διαφορετικούς τομείς όπως της υγείας, του εμπορίου, την οικονομική συνιστόσα αλλά και την προστασία των καταναλωτών. Έτσι λοιπόν και ο στόχος αλλά και η επιλογή των διαφορών ζημάτων που θα μας απασχολήσουν θα πρέπει να οδεύουν προς την προστασία των καταναλωτών αλλά και την απλούστευση των διαδικασιών που συνδέονται με τις νέες ίνες και τα νέα εφάσματα. Ένα στοιχείο που ενώνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επιχειρηματίες είναι ακριβώς ένας κοινός στόχος και η οικονομική διάσταση του ζητήματο. Το να αποσπάσουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα για την οικολογική επισήμανση είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Εμεί στην Ιταλία δεν το έχουμε προβλέψει αυτό. Στι διάφορε ετικέτε οφείλουμε στην Ιταλία να μιλάμε για την συντήρηση του ίδιου του προϊόντο με, ε, με διάφορα εικονογράμματα. Τα εικονογράμματα αυτά δεν πληρώνονται. Δηλαδή, κάθε χώρα, κάθε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαχειρίζεται αυτόνομα το σύστημα αυτών των εικονογραμμάτων. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που θα πρέπει να μα απασχολήσει. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μια σχετική ομοιομορφία. Ακόμα και για την περίπτωση του care labeling. Τα κόστη δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Δηλαδή, βάσει μελετών στην Ιταλία δεν ε, επιβαρύνει το και labeling ιδιαίτερα, διότι η ποσόστοση των ενώσεων, εφόσον κανείς αποτελεί μέρος κάποιες ένωση που έχει να κάνει με τα κλώστρα ή φαντουργικά, σημαίνει την δωρεάν παροχή αυτών των εικονογραμμάτων. Η δεύτερη πτυχή είναι μια εξίσου σημαντική πτυχή, η οποία συνδέεται με την ασφάλεια και τη χρήση των ουσιών στα υφάσματα. Δηλαδή, εδώ ερχόμαστε σε ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, το θέμα του REACH. Να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη το REACH είναι μια υποχρέωση. Πρέπει να σεβαστούμε τις προδιαγραφές που προκύπτουν. Αλλά αυτό όχι για τα εφάσματα και τα κλωστέφαντουργικά προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν η αρχή, η αρχή αυτή του REACH διατομεακά να ισχύει, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά και για αυτά που προέρχονται από την Κίνα. Σε μια φάση λοιπόν που τα προϊόντα αυτά μπαίνουν στην Ευρώπη ελεύθερα, θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική αυστηρότητα, ε, ε, μια πυγμή στο να ε, μπλοκάρουμε τα προϊόντα που ενδεχομένω δεν σέβονται τι προδιαγραφέ του REACH. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά σε πολλά κράτη κράτη που δεν υπάρχει ακόμη επαρκής ε, παρακολούθηση των αρχών του ΡΙΤΣ. Ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα προσφυλές στο έθνος μου, στην χώρα μου, είναι το ΜΕΝΤΙΝ. Προστασία των καταναλωτών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων, των βιοτεχνιών που εντοπίζουν την έννοια της ποιότητας, της ασφάλειας, στις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι όπως είπε μια συνάδελφος, η κυρία Μοσκαρντίνη, που από χρόνια ασχολείται με τα θέματα αυτά, έχει εργαστεί και ως νομοθέτης εδώ στη Ευρωκοινοβούλια για τα θέματα αυτά του Μεντίν, ε, ξέρει και εκείνη ότι υπάρχουν πολλά δυσκολία, πολλές δυσκολίες εδώ. Είναι ένα θέμα λοιπόν το μεντίν και το τελικό προϊόν. Αν ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο και στα εφαντουργικά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι τα εφαντουργικά, τα ενδύματα μπορεί να ξεφύγουν από την ευρεία αυτή έννοια του μεντίν η οποία έχει παραμείνει μπλοκαρισμένη σε επίπεδο από τέσσερα χρόνια. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα και τη χώρα προέλευσης σε όλες τις περιπτώσεις ε, για την Ιταλία, για το ε, κατά πόσον θα ασχοληθούμε με το φερμοάρι, το κουμπί, τα επιμέρους στοιχεία του ενδύματος ή το από πού προέρχεται το ύφασμα ή το ίδιο το ένδυμα. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει για το κάθε ένδυμα να θεωρήσουμε ότι το ύφασμα είναι το καθοριστικό στοιχείο για να ορίσουμε το μεντίν. Ο ορισμός, ο πλήρης ορισμός του Made in σημαίνει ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το προϊόν παράχθη και ε, συναρμολογήθηκε λίγο πολύ εντός του κράτους από το οποίο προέρχεται το ύφασμα. Αυτό όμως θα δημιουργήσει προβλήματα και στις επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει, έχουν οργανώσει την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες των δραστηριοτήτων τους και το Made in είναι αδύνατο να το πιστεί κατά 100%. Όμω ένα αρχικό στάδιο θα ήταν τουλάχιστον να αξιολογούμε την προέλευση των υφασμάτων. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Εδώ τώρα για τα μεγέθη. Ανακάλυψα ένα στοιχείο που το θεωρώ πολύ παράξενο. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόμουν στην Ιταλία και μιλούσα με μια υπεύθυνη που μου έλεγε ότι τα μεγέθη, ιδίω τα γυναικεία ρούχα, αλλάζουν ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε περίοδο κρίση ή όχι. Ε, οικονομικής ανάκαμψης δηλαδή. Στην περίοδο κρίσης το 40 μπορεί να γίνει 42, ενώ στην περίοδο ανάκαμψης το 42 θα γίνει 40. Σας ομολογώ ότι αυτό επαληθεύεται και στην πράξη, διότι εμείς οι γυναίκες τον αγοράζουμε ένα ρούχο, ε, διαπιστώνουμε αμέσως ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. Ακόμα και οίκοι μόδας, ιδιαίτερα σημαντικοί και γνωστοί, κάνουν χρήση αυτού του, αυτής της έννοιας και το χρησιμοποιούν και ως όπλο μάρκετινγκ. Δηλαδή, μια γυναίκα θέλει να αισθάνεται ότι είναι αδύνατη, ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση και προτιμά να αγοράσει το 40 42. Είναι αστείο λίγο, αλλά και παράξενο και πολύ κοινό μάλιστα και συμβαίνει στην πράξη. Οπότε το size labeling, η επισήμανση του μεγέθους θα ε, εξελιχθεί σε μάχη, ακόμα και από την άποψη της, ε, του marketing των διαφόρων εταιριών. Τώρα, για την επισήμανση, την πολλαπλή επισήμανση. Σαφώς δεν μπορεί να είναι πάπυρος, ούτε περγαμηνή, ούτε κυκλοπαίδεια η ετικέτα. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι δεν μπορούν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χειριστούν τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο να ομοιογενοποιήσουμε τις ετικέτες σε όλες τις χώρες. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να διατηρήσουμε την πολυγλωσσική διάσταση, αλλά να μπορεί να κοπεί η ετικέτα με τρόπο εύκολο εάν ενοχλεί τους καταναλωτές το μεγεθός της. Οπότε κάποτε στα προϊόντα θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται όλες οι ουσίες που μπορεί να συμπεριλαμβάνει το ύφασμα, αλλεργογόνα και ούτω καθεξής. Να τα διαβάζει ο καταναλωτής στη στιγμή της αγοράς του προϊόντος, να ενημερώνεται και μετά να τη βγάζει την ετικέτα. Και θα θυμάστε ότι στα παντελόνια σας κύριε Μάντερς κάποτε όταν ενοχλούσε η ετικέτα στο κάθισμα μπορούσατε να την βγάλετε. Να λοιπόν τι θέλουμε να επαναφέρουμε. Οι προτάσεις που λάβαμε τώρα από τις ενώσεις καταναλωτών είναι αυτές που βλέπετε πάρα πολύ χρήσιμες και θα ευχαριστήσω κιόλας για τα δεδομένα αυτά τους συνεισφέροντες <clears throat> Και είναι και ένα πολύ καλό κίνητρο αυτό, ένα κίνητρο για να πάμε λίγο παραπέρα από όσα μας ζητά ενδεχομένως η Επιτροπή. Δηλαδή να ασχοληθούμε μόνο με τις νέες ίνες. Υπάρχουν τομείς σημαντικοί που κινούν την οικονομία μας εδώ και Νομίζουμε ότι είναι και τα κομμάτια αυτά της αγοράς που βρίσκονται πιο κοντά στον καταναλωτή. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή εξήγηση, αν και σε δύο εβδομάδες θα προσέλθετε και στην Ιταλία για να επισκεφτούμε τον βιομηχανικό αυτό τομέα. Ευχαριστώ. Um, Εμεί ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ ζωηρή και δυναμική συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία κανείς θα μπορούσε να σχολιάσει, όμως θέλω να ξεκινήσω αναφέροντάς σας ότι κατά τη γνώμη μου η γνήσια πρόταση, η πραγματική πρόταση δεν είναι αυτή που μας δημιουργεί τώρα τα προβλήματα. Φυσικά και κάθε κίνηση διευκόλυνση αγορά είναι ευπρόσδεκτη και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει το πεδίο εφαρμογή της πρότασης να διευρυνθεί. Και να μπορέσουμε να καλύψουμε και την ετικετοθεσία. Συμφωνούμε με όλα αυτά. Το ζήτημα είναι κατά πόσον μπορούμε να βρούμε την πιο δόκιμη λύση. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα ε, είδος ρουχισμού να μπορεί να διαβάσει τη γλώσσα του από τι ύφασμα είναι φτιαγμένο. Εντάξει, δεν τι εταιρείε σχετικά με μια μακρά λίστα με διαφορετικέ γλώσσε, αλλά αν έχει κανένα μια τεράστια ετικέτα μέσα στο, στο, στη φόρα του, του ρούχου του, θα, θα το κόψει, οπότε δεν θα την έχει. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε όλες, όλες τις γλώσσες σε αυτή την ετικέτα. Θα πρέπει εμείς σαν αφετηρία να κάνουμε να σκεφτούμε τι είναι το πιο καλό για τον καταναλωτή. Ο οποίο να μπορεί στη γλώσσα του να διαβάσει αυτά τα οποία θέλει να πληροφορία. Ταυτόχρονα έχουμε τώρα καινούργια υφάσματα, καινούργιες ίνες, καινούργιες περιγραφές που μπαίνουν στην αγορά. Θα πρέπει επομένω να κάτσουμε και να εναρμονίσουμε την ορολογία ούτως ώστε να έχουμε την, την ίδια ονομασία ε, για κάθε χώρα. Αυτό γίνεται τώρα. Η εναρμόνιση της ορολογίας για τα παλιότερα υλικά είναι πιο δύσκολο. Και θα πρέπει αυτό να επιβληθεί ως υποχρεωτική ρύθμιση. Όπως ακριβώς και οι οδηγίες για το πώς πλένεται το κάθε ρούχο. Θα πρέπει επομένω να ενεργούν σύνομα όλοι αυτοί που παράγουν τέτοια προϊόντα. Γιατί πολλές φορές προβλήματα ανακύπτουν από λάθο οδηγίες. Λέει, πούμε, μόνο στεγνό καθάρισμα ή λέει μόνο πλήσιμο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό αναφέρεται από τον παραγωγό ε, ε, ε, ενώ έχει περιθώριο να πληθεί και αλλιώς το συγκεκριμένο ρούχο. Άρα, επομένως, θα πρέπει να φροντίσουμε να τηρούν την νομοθεσία η παραγωγή. Πολύ σημαντικό. Και αν έχουμε κάποια κατάλοιπα, κάποιες χημικές ουσίες επικίνδυνες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των ε, ρούχων, των υφασμάτων, θα πρέπει αυτό επίσης να το ξέρει ο Για τα μεγέθη τώρα. Καλό είναι να το ρυθμίσουμε και αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο θέμα. Στη Δανία χρησιμοποιούμε τα νούμερα που χρησιμοποιεί και η υπόλοιπη Ευρώπη. Καλά, εγώ το λεφτό που φοράω 36, αλλά είναι αγορισμένο στην Ιταλία. Και θα ε, λεγόταν 42, ε, αν δεν ήταν από την Ιταλία. Και αν ήταν 44, αυτό θα ήταν ντροπή, θα το παρά μεγάλο. Επομένως, ίσως είναι σωστή ιδέα να εναρμονίσουμε και τα μεγέθη. Αν λέμε ότι είναι νούμερο 42, θα πρέπει αυτό να το σε συγκεκριμένες απαιτήσει ε, μεγέθους. Αν θέλουμε οι καταναλωτές να αγοράζουν στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να στηριχτούν, να βασιστούν στο μέγεθος το οποίο ε, το οποίο τους λέμε. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει με την εποχή το μέγεθος. Αυτά όσον αφορά την εντολή που αφορά την οδηγία. Πολύ χρήσιμο αυτό και ίσως έτσι μπορούμε να κάνουμε κάτι και για τα μεγέθη. Και μην, υπάρχει, ε, μην υπάρχουν λάθη όταν έρθει η ώρα να αγοράσει ρούχο πριν την κυρία Ρουλέ. Για να δούμε λέει ο πρόεδρος τι είχε ετοιμάσει η γραμματεία εδώ πέρα της ε, Μόνιμης Επιτροπής για την ε, προτυποποίηση. Έχει εδώ πέρα ένα συγκριτικό πίνακα για όλα τα μεγέθη, για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Όλα αυτά θα σας τα μοιράσω. Έχει γίνει αυτή η δουλειά και είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένη και πλήρης. Σας υπενθυμίζω συνάδελφοι μιλούμε για αυτό το σχέδιο κειμένο που αφορά τα εφάσματα και όχι συγκεκριμένα διαρροχισμό. Γιατί τα διαρροχισμό μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά υλικά, οπότε υπενθυμίζω στην εισηγήτρια ότι θέλω να μας πείτε κάτι για, τα, για υφάσματα, ε, ονομασίες και μεγέθη. Γιατί κατόπιν ο κατασκευαστή ο παραγωγός αποφασίζει τι θα κάνει, πώ θα το ονομάσει. Αυτός που έχει μεταποιήσει το, το ύφασμα την πρώτη ύλη και έχει βγάλει ό,τι έχει βγάλει. Άρα προσοχή εδώ συνάδελφοι. Δεν λέω στο μέλλον να μην ασχοληθούμε και με τα ρούχα. Αλλά αυτή η πρόταση αφορά τα υφάσματα. Ακριβώς αυτό ήθελα και εγώ να πω, Πρόεδρε. Από το στόμα μου το πήρατε. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η έκθεση... Χάνομαι λίγο σε αυτή την έκθεση. Βεβαίω ενδιαφέρομαι για την Ιταλική βιομηχανία εγώ και γνωρίζω τα προβλήματά σας. Και στην πρωτοβουλία μου προσπάθησα όντω να συνδέσω και αυτό το θέμα του Made in. Αλλά δεν έχει χαθεί, πιστεύω, τίποτα. Και είμαι τη άποψη ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που υπάρχει εδώ, γιατί μιλούμε για το μέλλον της ε, βιομηχανίας και για τον bridge επίσης και με το θέμα των, ε, της προστασίας των δεδομένων, γιατί εκεί μιλούμε για πολύ περίπλοκες συζητήσεις. Πραγματικά λοιπόν θα σας ζητούσα επιγόντως να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα καθαρό κείμενο και να μην ατέρμο να συζητούμε για το ίδιο πράγμα, γιατί Αλλιώ θα μπορούσαμε να δούμε γιατί, θα μπορούσαμε να θέσουμε και το γιατί πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Κύριε Σβάμπ, και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μάντερ για να ανακεφαλαίωσει. Κύριε Ρόιτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η κυρία Ρούλα ακριβώς είπε αυτό που ήθελα και εγώ να πω. Θα ήθελα να δούμε το θέμα της επισήμανσης και θα ήθελα να πω ότι τα, α, οι άνθρωποι από τον τομέα της ε, υφασματοβιομηχανίας ε, πραγματικά ανησυχούν πολύ για, το, για τις ετικέτες για τις υποχρεωτικές ετικέτες, όχι μόνο για τους κατασκευαστές, αλλά και για τους πολιτές. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν ίσως να υπάρχουν ε, κάποιες προειδοποιήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, ε, ο κλάδος μας είπε ότι όντως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Οι εισαγωγείς πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια και η επισήμανση θα πρέπει να βοηθά την εφαρμογή του bridge Κύριε συνάδελφε, Μιλήσατε και για την ε, επισήμανση της χώρας προέλευσης. Αυτό ακούγεται εύκολο, αλλά εδώ και καιρό ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Αυτό σημαίνει τι ποσοστό της 100 του προϊόντος προέρχεται από ποια χώρα, για να μπορέσουμε να το ε, επισημάνουμε κιόλα. Ίσως αν υπήρχε μία ετικέτα με ευρωπαϊκή να μπορούσε να βοηθήσει τους κατασκευαστές, τους παραγωγούς και μετά να καθορίσουμε ας πούμε κάποια ποσοστά, ας πούμε 60%. Ότι, αυτό, ότι 60% θα πρέπει να προέρχεται από την Ευρώπη, ας πούμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά υφάσματα, εισάγουμε πάρα πολλά υφάσματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ε, συγκεκριμένες ε, μάρκες ε, οι οποίες παράγουν τα συγκεκριμένα υφάσματα και όλοι ράβουν τα υφάσματα και τα ρούχα τους στην Ασία. Επομένως, τι ετικέτα θα βάλουμε made in. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξηγήσουμε και στους καταναλωτές. Πρέπει να το ξέρουν αυτό οι καταναλωτές, ότι τα υφάσματα που φορούν είναι ασφαλή από πλευράς υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ασχολούμαστε με τα μεγέθη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μπούμε στην ουσία του κανονισμού. με την νέα αυτή πρόταση οι διαφορές νομίζω θα... Ο νέος κανονισμός θα βελτιωθεί με αυτές τις νέες ίνες που προτείνονται. Θα μπορέσουμε να ε, άρουμε κάποιες επιφυλάξεις των κρατών μελών και να προωθήσουμε τις αγορές τους. Βέβαια αυτή η εισαγωγή των ε, καινοτόμων νέων ινών θα πρέπει να προωθηθεί θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και στον κανονισμό, στο σημείο που μιλά για την καινοτομία στην εσωτερική αγορά. Φυσικά υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία είναι αρκετά ακαθόδη, ε, επισήμανση στα, των μεγεθών, ε, πτυχές υγείας κτλ. Ε, μιλούσαμε και για την εργασία παιδιών, για την κατασκευή αυτών των υφασμάτων. Και επίσης με αυτά τα θέματα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Στο σχέδιο του κανονισμού βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά από αυτόν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θέλουμε ένα ευέλικτο και ανάλογο σύστημα ρυθμίσεων για τον τομέα της κλωστοφοντουργίας. θα μπορούσε να είναι ε, ε, επιτρεπτό για όσους το επιθυμούν σε ό,τι αφορά την επισήμανση. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία υποχρεωτικά στις ετικέτες. Το ίδιο ισχύει και για τα μεγέθη. Το πρότυπο που προτείνεις Μάλκομ Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να, να εφαρμοστεί. Εγώ φοράω νούμερο 40, ας πούμε. Δεν ξέρω σε σχέση με, αυτά... με τα ρούχα της κυρίας Μόζε τι μέγεθο είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ε, καλή επιτυχία στον εισηγητή για την ε, περαιτέρω επεξεργασία της έκθεσης του. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα μεγέθη. η Επιτροπή να απαντήσει. Ευχαριστώ. Μιλούμε εδώ για απλούστευση, Πρόεδρε. Η Κομισιόν προτείνει αυτόν τον οικονομισμό για να απλουστεύσει τον, το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Κομισιόν είναι ανοιχτή σε συζήτηση για οποιαδήποτε άλλη πτυχή περί επισήμανσης, αλλά θα ήθελα να το κάνουμε αυτό ξεχωριστά από την πρόταση που βρίσκεται εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα άμεσα. Και εμείς καλωσορίζουμε την μελέτη και τις πληροφορίες που μας παρέχει και βεβαίως την περιμένουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω. Αν ενδιαφέρεστε, θα μπορούσα να σας δώσω μια σύντομη ενημέρωση των εργασιών στο Συμβούλιο. Έχουμε ε, ασχοληθεί με τα κράτη-μέλη αρκετά αποτελεσματικά με το θέμα αυτό και η Σουηδική Προεδρία και η Κομισιόν θεωρεί ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ε, συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Το νέο κείμενο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουν συζητήσεις με το Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν. Η βασική διαφορά ίσως να είναι η εισαγωγή κάποιων αναφορών στην τυποποίηση σε ό,τι αφορά τι μεθόδου στο παράρτημα 8 που είναι πολύ τεχνικό. Και για τα υπόλοιπα είναι κάποιες τεχνικές αλλαγέ που πρέπει να γίνουν για να ε, υπάρξει καλύτερη σαφήνεια του κειμένου και ασφάλεια δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ζήτημα που θέσατε για το πεδίο της οδηγίας αυτής είναι ακριβώς και το αντικείμενο της συζήτησης όταν συναντηθήκαμε με τους κοιόδης εισηγητές. Θα αντιγράψουμε πιστά το πεδίο όπως μας προτάθηκε, γιατί εξ όσων κατάλαβα εγώ, δεν είχε τόσο αρνητικέ πτυχέ η πρόταση τη Επιτροπή όπω την ε, είδαμε μέσα από τη συζήτησή μα. Όμω και η ομάδα εργασία των εισηγητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τα πράγματα για του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Εάν λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το πράξουμε. Θα πρέπει να διευρύνουμε όμω το πεδίο. Αυτό ήταν το συμπέρασμα τη συνάντηση με του σχεώδει εισηγητέ. Επίση, συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουν και εκείνοι τι πλέον εκτίματα θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε. Θέλουν να επιταχύνουμε παράλληλα τη διαδικασία. Να επιταχύνουμε λοιπόν, να συμφωνήσουμε αυτή τη στιγμή με το κείμενο που έχουμε απειτάπητο και στο μέλλον θέτουμε και νέε προτάσει για την επισήμανση. Εάν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με σκοπό την βελτίωση των ετικετών τη επισήμανση, ίσω ήδη αυτό είναι αρκετό. Όμω και πάλι θα πρέπει να έχουμε πληροφορίε, επαρκεί πληροφορίε για να δούμε την εφικτό, τι μπορούμε να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πολίτες, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα για την όλη διαδικασία ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τελευταίο συμπέρασμα ίσως είναι ότι ας δούμε το πεδίο και μετά με τις γνώσεις που έχουμε και τη συνδρομή της Επιτροπής Ίσως, ίσως ε, η ακριβή συνδικαιτοθεσία όπως θα την προτείνουμε εμείς να συζητηθεί και να υποβληθεί και ως νομοθετική πρόταση. Όμως ως πολιτικοί θύνοντες να λάβουμε κάθε ευκαιρία που μας προσφέρεται για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο ιδίως προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και την οικονομία. Αν βελτιώσουμε λοιπόν εδώ τα πράγματα νομίζω ότι θα έχουμε κάνει τη δουλειά μας πολύ καλά. Όπως άλλωστε προβλέπουν και οι υποχρεώσεις μας ως εκλεγμένων εκπροσώπων των πολιτών. Από τεχνικής λοιπόν άποψης η πρόταση είναι αρκετά περίπλοκη, αλλά ε, εάν διευρύνουμε το πεδίο θα γίνει ακόμη πιο περίπλοκη όσο ακριβώς εμείς θέλουμε. Στο τέλος νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια ισορροπία και συμβαστικές προτάσεις και σε ό,τι αφορά το Made μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα στην μήνυ Ολομέλεια η Επιτροπή θα απευθύνει δήλωση για, για το θέμα αυτό του Made Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα τότε. Και στο τέλος νομίζω ότι θα έχουμε μια ισορροπή και πραγματικά χρήσιμη έκθεση. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάντερς. Ως προς το χρονοδιάγραμμα τώρα. Τι προβλέπετε. Περιμένετε το χρονοδιάγραμμα, περιμένετε μάλλον να ολοκληρωθεί η μελέτη, γιατί όπως ξέρουμε εγκρίθηκε από τους συντονιστές και ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά δεν είμαι βεβαίω πώ ακριβώ θα εξελιχθεί χρονικά. Έχετε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για το τι προτείνετε και πότε θα έχετε καταλήξει μια πρώτη πρόταση. Ναι. Το δικό μου συμπέρασμα ήταν ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε περί τίνος συζητάμε, γιατί ωραία είναι να μιλάμε στο βρόντο, αλλά χωρίς ειδικέ γνώσεις αυτό δεν γίνεται. Το συμπέρασμα της συνάντησης με τους συντονιστές τους εισηγητές, συγγνώμη, τους σκεώδεις εισηγητές, ήταν να περιμένουμε μέχρι να αποφανθούν οι ειδικοί της μελέτη. Όπω άκουσα και από την γραμματεία θα γίνει αυτό στι αρχές Ιανουαρίου. Τότε μπορούμε να επιταχύνουμε και να ψηφίσουμε ενδεχομένω το Μάρτιο, στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Νομίζω ότι είναι καλό ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Το συμφωνήσαμε λίγο πολύ και αν θέλετε μπορούμε ήδη να σας δώσουμε το χρονοδιάγραμμα, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε διαβάσει τη μελέτη. Ανυπομονούμε. Προφανώς έχετε χρονοδιάγραμμα και για τη μελέτη, οπότε περιμένουμε τα πορίσματα της μελέτης αυτής και της ε, ανεπίσημης επισκέψής σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερως. Ε, κυρίε και κύριοι, κλείνουμε τώρα τι εργασίε τη Επιτροπή μα. Για απόψε το βράδυ θα έχουμε και κλεισμένο των θηρών μια συνέντευξη των συντονιστών και ο κύριο Μπέναν από τη Γενική Διεύθυνση Αγορά θα μιλήσει στου συντονιστέ για ένα ζήτημα που εγέρθη ε, σε σχέση με τη διαδικασία τη επιτροπολογία. Προσκαλώ λοιπόν όλου του υπόλοιπου πέραν των συντονιστών και όσων έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη συνάντηση αυτή να αποχωρήσουν για να περάσουμε στο επόμενο μέρος της συνάντησης σας περιμένω αύριο στις 9 για την τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας με πολλά σημαντικά θέματα επιτάπητος όπως την αναθεώρηση των βιοκτώνων προϊόντων και τους σχετικούς κανόνες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη μέχρι τώρα συμμετοχή τους.